Ε, Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, καλώ ήρθατε. Θα αναλάβω την Προεδρία της Επιτροπής μας εν μέρη, διότι ο Πρόεδρος μας είναι λίγο αδιάθετος. Πρέπει να μείνει ακίνητος, οπότε περιμένοντάς τον θα προεδρεύσουμε εγώ και η συνάδελφος, η κυρία Ντελβό, εάν θέλει. Εναλλασσόμενη. Ωραία. Μερικές ανακοινώσει αν μου επιτρέπετε. ώστε να πάρει και την τελική τη μορφή μερική διάταξη. Πρώτα απ' όλα σημειώστε ότι το σημείο 9 θα εξεταστεί μετά το 7. Το 2 θα συζητηθεί μετά το 9. Το 5 μετά το 12. Το 20 και το 21 θα συζητηθούν μετά το 15. Τα λέω όσο μπορώ πιο αργά για να προλάβετε να σημειώσετε. Δεν είναι απλό να παρακολουθεί κανείς όπως είπε η κυρία Ντελβό, αλλά κάνω ό,τι μπορώ. Ε, το 23 μετά το 13, το 28 και το 29 μετά το 31 και εν τέλει το 30 μετά το 26. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, συμφωνούν όλοι. Σας ευχαριστώ. Αποφασίστηκε λοιπόν. Να σας πω καταρχάς ότι ο κύριος Μαστάλκα δεν μπορεί να μετακινηθεί επειδή υπέστη χειρουργική επέμβαση και στην Επιτροπή μας θα τον αντικαταστήσει η κυρία Μάλιν Διόρκ, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα. Μάλλον ναι, είναι εδώ, τη χαιρετούμε. Καλώς ήρθατε. Κατά τα άλλα, να σας ε, επισημάνω ότι μετά τη συνεδρίαση της 5ης Σεπτεμβρίου, οι συντονιστές ο κύριος Μπερνάρ Μονό υπέβαλε έκθεση για τον κανονισμό 133, για, τον, για το άρθρο 133 του εσωτερικού κανονισμού σε σχέση με τους κανόνες του, του, κάτι δεν πάει καλά με τις σημειώσεις μου, με τους κανόνες του για την πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα δύο πρώην Ευρωπαίων Επιτρόπων. Θα ξέρετε ποιοι είναι, γιατί θα τα διαβάσατε πρόσφατα και στον τύπο. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης. Με συγχωρείτε, θα μου περάσει σε πέντε λεπτά, θα συνηθίσω. 13 και 14 Ιουνίου 2016. Έχετε αντιρρήσεις για τα πρακτικά. Εφόσον αντικατοπτρίζω συζητήθηκαν εκεί, εγκρίνεται ολοσχερός και τελεσιδίκος. Πριν περάσουμε στο ζουμί της ε, συζήτησής μας σήμερα, της συνεδρίασης, να σας χαιρετήσω συνάδελφοι, διότι προστεθήκατε στο μακρύ κατάλογο των Γάλλων ε, φορολογουμένων που θα έχετε, που μόλις αποκτήσατε ένα παιδί. Ε, σας συγχαίρουμε για το μωρό. Ε, με τόσο μεγάλη λοιπόν ε, χαρά και ευχάριστη διάθεση να περάσουμε στην ουσία της συζήτησής μας. Ο κύριος Σάγερ. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο, ένα λεπτάκι μόνο. Να θυμίσω στους συναδέλφους ότι πριν από μισό περίπου χρόνο, πέντε μήνες δηλαδή, η Επιτροπή μας ε, συμφώνησε να πάρει μέρος σε μια διαδικασία κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα κατεπήγον διαδικαστικό εδώ στο Κοινοβούλιο όπου ομόφωνα, με δύο αποχές μόνο, αποφασίσαμε να ζητήσουμε από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου να κοινοποιήσει στο Συμβούλιο το γεγονό ότι είμαστε δεσμευτημένοι με τη διαδικασία του περασμένου Σεπτεμβρίου. Κατεπίγουσα διαδικασία για την υποχρεωτική κατανομή των προσφύγων. Θεωρήσαμε ότι δεν ε, συνεισέφερε επαρκώς την απόφαση το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή μας δεν μελέτησε το θέμα όσο θα θέλαμε και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να το κοινοποιήσουμε στο Συμβούλιο. Στα πλαίσια των έκτακτων ε, διαδικασιών, λοιπόν, τέτοιου είδου ε, πρακτικέ δεν μπορούμε να τι δεχτούμε και στο μέλλον. Ε, και ανησυχώ γιατί δεν είδα κανένα ίχνο αυτή τη κοινοποίηση πέραν τη επιστολή του Πρόεδρου Σούλτ. Δεν ανελήφθη καμία δράση και πιστεύω ότι η Επιτροπή μα θεωρεί ότι οι συζητήσει εδώ είναι πολύ σοβαρέ και θα έπρεπε να έχουν κάποια επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα. Θα θέλαμε λοιπόν, Πρόεδρε, να ρωτήσετε τον Πρόεδρο Σούλτς αν σκοπεύει να κοινοποιήσει και να ενημερώσει το Συμβούλιο για τις μέριμνές της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ κύριε Σάγερ. Καταγράφουμε την ε, ε, δική σας την ε, παρατήρηση και προχωρούμε. Να καλωσορίσουμε την κυρία Μάρτα Περτεγκάς, η οποία είναι διευθύντρια ε, του μόνιμου γραφείου της συνδιάσκεψης της Χαϊκής για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Έχετε το λόγο. Πού βρίσκεστε? Ωραία. Ευχαριστώ και καλό απόγευμα. Κυρίε και κύριοι, εξωτερικά μέλη του Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι άλλων θεσμικών οργάνων της Ένωσης, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να σας παρουσιάσω σήμερα ένα από τα σχέδια προτεραιότητα τη οργάνωση που εκπροσωπώ εδώ, την διάσκεψη τη Χάιζερ του Διεθνέ Δίκαιο. Επειδή έχετε φορτωμένη μέσα διάταξη, θα αναρωτιέστε πώ αυτό συνάδει με τι εργασίε σα. Και βεβαίω, ε, επειδή είναι φορτωμένη μέσα στη διάταξή σα, ε, είναι κάπως δύσκολο να κάτσετε να σκεφτείτε τι κάνουμε εμείς. Όπως θα γνωρίζετε, είμαστε ένας ενεργός οργανισμός σε ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου. Έχουμε ένα πολύ ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων, μια σειρά από διεθνείς συμβάσεις ε, γνωστές ε, ε, για τις υιοθεσίες των παιδιών, μεταξύ άλλων και είμαι εδώ για να σας μιλήσω σήμερα για την πρόοδο των εργασιών μας έτσι ώστε ενδεχομένως νωρίτερα από ό,τι ε, περιμέναμε να γίνουμε μια νέα σύμβαση για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων από άλλη χώρα. Υπάρχει ήδη μια παρουσίαση, την οποία λογικά πρέπει να βλέπετε στην οθόνη. Τέσσερα σημεία είναι αυτά που οποία θέλω να επικεντρωθώ. Το θέμα αφενός τη σημασία του τομέα αυτού, δηλαδή αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων. Θα σας παρουσιάσω βεβαίως ε, αυτό το σχέδιο σχετικά με τις αποφάσεις και πού έχουμε φτάσει ως τώρα, ποιες είναι οι εξελίξεις. Πολύ σύντομα, ε, βεβαίως υπάρχουν πολύ περισσότερα στοιχεία στο PowerPoint, δεν θα μπω ε, στις λεπτομέρειες ε, σε ό,τι αφορά το σχέδιο ψηφίσματος για την Σύμβαση του 2016 το σχέδιο σύμβασης μάλλον και θα σας πω επίσης ε, πώς, τι, πώς έχει το κείμενο αυτή τη στιγμή και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Τι δηλαδή θα γίνει στο άμεσο μέλλον έτσι ώστε να μπορέσει να συναυθεί αυτή η σύμβαση. Όπως θα γνωρίζετε, η σύμβαση της Χάγης δεν διεκδικεί την αποκλειστικότητα σε ό,τι αφορά την αναγνώση και την εκτέλεση των ξένων αποφάσεων και στο εθνικό δίκαιο υπάρχουν ε, σχετικές διατάξεις Υπάρχει λοιπόν το θέμα κατά πόσο μια τέτοια απόφαση θα έχει άμεση εκτέλεση, άμεση ισχύ ή θα πρέπει να υπάρχει μια διμερή συμφωνία για να συμβεί αυτό. Είναι διαφορετικές οι απαντήσεις που δίδονται στα εθνικά νομικά συστήματα καθώς ε, και στα πλαίσια των διμερών συμφωνιών που έχετε συνάψει με πολλές άλλες χώρες ανά τον κόσμο και βεβαίως ε, υπάρχουν και μια σειρά από διεθνή νομικά μέσα Επιτρέψτε μου εδώ ε, να αναφερθώ και στα ε, υπερεθνικά μέτρα, ε, μέσα μάλλον, όπως η Σύμβαση των Βρυξελών 2B. Υπάρχει λοιπόν ο κανονισμός Βρυξέλλες 1. Υπάρχουν, υπάρχουν μια σειρά από διεθνείς συνθήκες από το 1967 για το ζήτημα της εκτέλεσης και της αναγνώρισης. Γιατί λοιπόν χρειάζεται μια σύμβαση. Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα. Γιατί η, η οργάνωσή μας εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή. Φανταστείτε μια απόφαση που έχει παθεί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που πρέπει να εκτελεστεί στην Κίνα ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επειδή παραδείγματος χάρη τα περιουσιακά αγαθά της εταιρεία που έχει χάσει τη δίκη βρίσκονται εκεί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο εφαρμοστέο νομικό μέσο για αυτές τις, για αυτές τις περιπτώσεις. Μπορεί να υπάρχει βεβαίως μια διμερής ε, συμφωνία με την χώρα, την εν λόγω χώρα. Αλλά σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο γενικά εφαρμοστέο νομικό μέσο. Αυτό είναι το κενό που θα πρέπει να καλύψουμε. Πρόκειται για ένα σχέδιο τη διεθνού νομική κοινότητα εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες ένα ζήτημα λοιπόν που επανέρχεται στην μέση διάταξη των εργασιών μα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Θα μπορούσα βεβαίω να αναφερθώ στο τι είναι μέχρι και πριν από 100 χρόνια. Αλλά νομίζω ότι σα ενδιαφέρει πιο πολύ το σήμερα. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Χάγη και, και τι πρέπει να γίνει για να τα καταφέρουμε. Αυτά για το ιστορικό να σας πω ότι το σχέδιο των αποφάσεων έτσι όπως το γνωρίζουμε ξεκίνησε το 1992 που είναι το έτος που εγώ ολοκλήρωσα τις νομικές μου σπουδές στη Βαρκελόνη πριν από αρκετό καιρό δηλαδή όπως αντιλαμβάνεστε Πρόκειται λοιπόν για ένα μακροσκελές σχέδιο σε τρεις φάσεις θα μπορούσαμε να πούμε. Η αρχική φάση από το 1992 στο 2001 εδώ η ιδέα ήταν, να χρησιμοποιήσω αυτούς τους όρους αν μου επιτρέπετε, να μπορέσουμε να επαναλάβουμε σε παγκόσμιο επίπεδο ένα εξαιρετικά επιτυχές μοντέλο που υπάρχει στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει στην Ευρώπη δικαιοδοσία και για την αναγνώριση και για την εκτέλεση, δηλαδή ποιο αποφασίζει, πού αποφασίζεται κάτι τέτοιο, είναι ένα μοντέλο το οποίο λειτουργήσε σωστά στην Ευρώπη από το 1968 χάρη στη Σύμβαση των Βρυξελών. Ήταν λοιπόν ένα μοντέλο το οποίο θέλησαμε να αναπαράγουμε. Είχαμε μια σειρά από νομικά μέσα. Ένα από αυτά είναι το κείμενο του 2001. Δυστυχώς όμως δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία η όλη διαδικασία, ίσως να ήταν υπερβολικά φιλόδοξο το εγχείρημα. Γι' αυτό λοιπόν η Σύμβαση της Χάγης, η οργάνωση την οποία εκπροσωπώ, αποφάσισε να επικεντρωθεί ε, σε κάτι πιο συγκεκριμένο. Να ασχοληθούμε δηλαδή με τα εμπορικά ζητήματα και πιο συγκεκριμένα με ζητήματα όπου έχουν αποφασίσει τα συμβαλόμενα μέρη ποιο δικαστήριο θα έχει διεθνή δικαιοδοσία. Ε, αυτό μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει μια επιλογή δικαστηρίου. Να υπάρχει μια συμφωνία για επιλογή δικαστηρίου. Μπορεί να γίνει και μέσω μια ε, συμφωνία διατησία. Υπάρχει ήδη γι' αυτό κάποιο νομικό καθεστώ, η Σύμβαση τη Νέα Υόρκη. Οπότε εδώ αυτό που θέλησαμε να κάνουμε είναι να δούμε τι θα κάνουμε αν αντί για διατησία ε, αποφασίσουμε να καθοριστεί εκ των προτέρων το δικαστήριο και όποια απόφαση να πάρει το δικαστήριο αυτό να μπορεί να εφαρμοστεί και να, να εκτελεστεί σύμφωνα με κάποιου κοινού κανόνε. Η απάντηση ήταν ναι, διότι το 2005 εγκρίθηκε η σύμβαση για την επιλογή του δικαστήριου και ε, τέθηκε σε ισχύ και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να βεβαίω να ευχαριστήσω την για την υποστήριξη ε, κατά την εφαρμογή της ε, σύμβασης τέθηκε σε ισχύ χάρη στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της σύμβασης αυτής και ξέρω ότι αυτή η Επιτροπή υποστήριξε ε, σε μεγάλο βαθμό το κείμενο αυτό, το νομικό μέσο αυτό έτσι ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επικυρώσει τη σύμβαση στη Χάγη. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή ενισχύ αυτή η συμφωνία, συμμετέχουν 29 χώρες, μια από αυτές τις χώρες είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και σε πέντε ημέρες θα, έχουμε, ε, θα φτάσουμε στο 30ο μέλος, τη Σιγκαπούρη. Αυτά για να σας δείξω ότι αυτή η φάση προχωράει καλά σε ό,τι αφορά τα, τις αποφάσεις, το σχέδιο για τις αποφάσεις. Τώρα από εκεί και πέρα είπαμε ότι η σύμβαση αυτή αφορά την επιλογή του δικαστηρίου, τις συμφωνίες για επιλογή δικαστηρίου μάλλον. Όμως υπάρχουν πολλών μορφών ε, διαφορές όπου δεν υπάρχει κάποια ρήτρα επιλογής δικαστηρίου. Τι γίνεται με τις αποφάσεις αυτές ε, θα έχουν κάποια ισχύ πέρα από τα, από τα σύνορα της χώρας όπου πάρθηκε απόφαση. Τέθηκε το ερώτημα σε μια ομάδα πυρογνωμόνων νωρίτερα και έχει αποτελέσει αντικείμενο εργασιών μιας ομάδας εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή της αρχή ήταν εξαιρετικά ενεργό μέλος τη ομάδα εργασία αυτή και εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην λόγω ομάδα εργασία, την οποία ευχαριστούμε ε, που βρίσκεται εδώ σήμερα και βεβαίως υπάρχει πολύ ενεργή παρέμβαση και ενδιαφέρον από πολλές ε, χώρες που εμπλέκουν στην διαπραγμάτευση. Βεβαίως πάντα το ερώτημα τι κάνουν οι Αμερικανοί έτσι. Οι Αμερικανοί δηλαδή είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν στον τομέα αυτόν. Είναι διατεθειμένοι να δεχθούν οι αποφάσεις ευρωπαϊκές να εφαρμόζονται και να αναγνωρίζονται στις ΗΠΑ. Για την ώρα η απάντηση είναι θετική. Υπάρχει ένα σχέδιο κειμένου το οποίο προετοίμασε η ομάδα εργασίας στο τέλος του 2015 και τώρα περνάμε στην επόμενη φάση, μια σημαντική φάση των εργασιών, η Ειδική Επιτροπή. Η Ειδική Επιτροπή ουσιαστικά ε, σημαίνει ότι συμμετέχουν όλες ε, οι χώρες ε, που εμπλέκονται στη σύμβαση αυτή, 81 χώρες πιο συγκεκριμένα, που ένα πολύ πιο ευρύ σχήμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η Επιτροπή εξετάζει το κείμενο που έχει προτείνει η ομάδα εργασία. Τον Ιούνιο συνήλθε για πρώτη φορά η Ειδική Επιτροπή και θα ξανασυνέλθει ε, τον Φεβρουάριο του χρόνου. Προχωρούν οι εργασίες, οπότε το θέμα βεβαίως από εκεί πέρα είναι πού έχουμε φτάσει Έως τώρα λοιπόν έχουμε το σχέδιο ε, σύμβασης το 2016 έχει και γραμματεία το έγγραφο και μπορείτε να το δείτε όποτε θέλετε. Θέλουμε λοιπόν να απαντήσουμε αφενός στο ερώτημα που έθεσα νωρίτερα, να εξασφαλίσουμε δηλαδή ότι όταν παίρνετε μία απόφαση σε οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης και πρέπει να ε, ε εκτελεστεί στο Μαρόκο ή στην Κίνα, να υπάρχουν απλοί, βέβαιοι και προλέψιμοι μηχανισμοί για να συμβεί αυτό. Και βέβαια αυτό είναι αμοιβαίο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι και οι αποφάσει που παίρνονται εκεί θα πρέπει να την χάνουν τη ίδια ε, τύχη εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου. Ακούστε, μιλήσατε 13 λεπτά, αν θέλετε μιλήστε άλλα 5. Προτιμώ να ρωτώ για να μην καταχαριστώ το χρόνο σας, του χρόνου σας. 5 λεπτά ακόμα λοιπόν και στη συνέχεια θα λάβετε μια παρουσίαση PowerPoint εφόσον το επιθυμείτε, εφόσον ενδιαφέρεστε. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του κειμένου συνοψίζονται λέγοντας ότι το παρόν εργαλείο, το παρόν μέσο, νομικό μέσο, δεν είναι όπως το προηγούμενο, που ήθελε να αντιμετωπίσει και το θέμα της διεθνούς δικαιοδοσίας και της αναγνώρισης και της εκτέλεσης. Εδώ ασχολούμαστε μόνο με την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων. Δεν μπαίνουν τα ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας που θα πρέπει να και κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα συμβαλόμενα μέρη που θα επικυρώσουν μια τέτοια συμφωνία. Δεν μιλάμε δηλαδή για διεθνή δικαιοδοσία. Μια άλλη ε, σημαντική διαφορά είναι ότι αυτό το μέσο δεν θα είναι το μόνο δεν θα είναι το μόνο πρότυπο αν θέλετε στον κόσμο. Μπορεί να υπάρξει αναγνώριση και εκτέλεση με βάση ε, την ε, εθνική νομοθεσία ή κάποιο περιφερειακό μέσο ή κάποια διμερή συμφωνία. Ε, εάν δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άλλοι κανόνες πιο ευνοϊκοί που να επιτρέπουν αναγνώριση και εκτέλεση πέρα από αυτά που προβλέπουμε εμείς εδώ, βεβαίως να τα εφαρμόσετε. Η σύμβαση όσο έχει αυτή τη στιγμή βασίζεται στη σύμβαση του 2005, δεν θα σας εκπλήξει αυτό, ήταν ένα επιτυχές εργαλείο, 30 συμβαλόμενα μέρη έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν θα σας κουράσω τώρα με διάφορες λεπτομέρειες για το πώς δηλαδή λειτουργεί αυτή η σύμβαση, καθώς και το πεδίο εφαρμογής της. ποια είναι η βάση για την αναγνώριση, για την εκτέλεση. Όπως μου ζητήθηκε θα αναφερθώ στο τι μας περιμένει στο μέλλον. Γιατί θεωρούμε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Είπαμε ότι το 1992 υπάρχει αυτό το σχέδιο για τις αποφάσεις την Σύμβαση της Χάγης. Γιατί λοιπόν είμαστε τώρα αισιόδοξοι, γιατί θεωρούμε ότι τώρα ενδεχομένως να μπορέσουμε να κλείσουμε επιτυχώς ε, το όλο εγχείρημα. Νομίζω ότι έχω απαντήσει στην πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα momentum, ε, μια θετική συγκυρία στις ενδιαφερόμενες ε, χώρες, όταν όλοι οι βασικοί εμπλεκόμενοι, η Κίνα, οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Σιγκαπούρη, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, όταν λοιπόν όλες αυτές οι χώρες προσέρχονται στο τραπέζι διαπραγματεύσεων θεωρώντας ότι είναι η στιγμή για μια συμφωνία, ε, είναι σημαντικό ε, να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο για να συμβεί αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα το τι μας λείπει, θα πρέπει την επόμενη φορά να επικεντρωθούμε στην επόμενη συνεδρία της Ειδικής Επιτροπής στις τελικές ρήτρε. Θα πρέπει δηλαδή να απαντήσουμε σε κάποια ερωτηματικά, σημαντικά ερωτήματα τη διάρθρωση με άλλα νομικά μέσα, μεταξύ των οποίων και οι Ευρωπαϊκέ Νομοθεσίε, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Αυτό ακόμα είναι μπροστά μα. Για να το πράξουμε αυτό και για να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο προ την τελική φάση τη Σύμβαση τη Χάγη. και ξέρω ότι κάθε οργάνωση έχει τι ιδιαιτερότητέ τη σε ό,τι αφορά την, τις διαδικασίες εργασίας. Εμείς ε, κλείνουμε με μια διπλωματική σύνοδο και ελπίζουμε αυτό να γίνει πριν το 2018 θα έχουμε λοιπόν και άλλες συζητήσεις έως ε, τότε. Το πιο σημαντικό όμως, και πρέπει να το υπογραμμίσω, είναι ότι το σκέλος που αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία δεν, είναι κάτι, δεν είναι κάτι που το έχουμε ξεχάσει. Όπως είπα νωρίτερα, σε μια προηγούμενη φάση, ο συνδυασμός της δικαιοδοσία και της αναγνώρισης και της εκτέλεσης σε ένα ενιαίο νομικό μέσο ήταν υπερβολικά φιλόδοξο, δηλαδή δεν τα καταφέραμε. Το Συμβούλιο όμω έχει, έχει ήδη συμφωνήσει ότι θα δημιουργηθεί μια ομάδα εμπειρογνωμόνων όταν ολοκληρωθεί το έργο τη Ειδική Επιτροπή και τότε θα εξετάσουμε κατά πόσο θα μπορούσαμε να έχουμε ένα νέο νομικό μέσο που θα αφορά τη δικαιοδοσία. Δεν είναι κάτι που το έχουμε ξεχάσει. Ε, θα επανέλθουμε και όταν ολοκληρώσει τι εργασίε η Ειδική Επιτροπή θα το δείτε. Τέλο, το 2018 Ελπίζουμε να έχουμε μια επιτυχή διπλωματική συνόδο, δηλαδή στη σύμβαση, για τη σύμβαση της Χάγης ε, θα μπορέσει να εγκριθεί αυτή η νέα σύμβαση. Ε, αυτά σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα. Ελπίζω να μάθατε κάτι. Είμαι στη διάθεσή για να απαντήσω οποιοδήποτε ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε για την ε, ευστοχία της παρουσίασής σας και τώρα να ακούσουμε την κυρία Βάντερκερ και από την Επιτροπή και μετά θα συζητήσουμε μαζί σας. Σας παρακαλώ να παραμείνετε εδώ για λίγο, γιατί μπορεί να χρειαστεί να ξαναπάρετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ την διευθύντρια του γραφείου που παρουσίασε το πρόγραμμα στην Επιτροπή σας. Πρέπει να σας πω ότι από την πλευρά της Επιτροπής είμαστε πολύ δραστήριοι σε όλο αυτό το πρόγραμμα και το στηρίζουμε. Η σύμβαση αυτή είναι ένα εργαλείο που το περιμέναμε εδώ και πολλά χρόνια στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Ένα πλαίσιο που θα επιτρέψει να έχουμε προβλεψιμότητα για το ιδιοσυναριακό εμπόριο και τις επενδύσεις. Για να καταλάβουμε καλύτερα ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος, πρέπει να το συγκρίνουμε με τον εσωτερικό μας ε, κανονισμό, τον κανονισμό Βρυξέλλες 1, ο οποίος ε, διευθετεί το θέμα των δικαιοδοσιών μεταξύ των κρατών μελών και προβλέπει ένα σύστημα για την αναγνώριση και την επιβολή δικαστικών αποφάσεων μεταξύ κρατών μελών. Η σύμβαση αυτή κάνει κάτι παρόμοιο, αν και όχι πανομοιότυπο, όπως μας εξήγησε η διευθύντρια του συνδιάσκεψης της Χάγης, σε σχέση με όσα συμβαίνουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντός λοιπόν Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε μια διπλή σύμβαση, δηλαδή και δικαιοδοσία και αναγνώριση και επιβολή και σε διεθνέ επίπεδο ξεκινάμε με την αναγνώριση και επιβολή, αλλά όπω ε, ακούσαμε Υπάρχει ένα λογικό χρονοδιάγραμμα για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αναγνώρισης επιβολής. Εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό είναι άκρο σημαντικό. Θα θυμάστε ότι όταν τα συζητήσαμε αυτά στην Επιτροπή σα, τα θέματα τη ε, αναδιατύπωση του κανονισμού Βρυξέλλε 1, με τον κύριο Ζεύκα τότε να προεδρεύει, Είχαμε ασχοληθεί με το πώ θα διαθετήσουμε και τι νομικέ μα σχέσει με τρίτα κράτη τότε και υπήρχε τότε η μέρημνα ότι καλύτερα θα ήταν να τα αντιμετωπίσουμε αυτά μέσω μια διεθνού σύμβαση. Η σύμβαση λοιπόν αυτό ε, αποζητά να κάνει. Είναι η συνέχεια που δόθηκε στην δική μα την αναδιατύπωση του κανονισμού Βρυξέλλες 1 πριν από μία διετία. Νομίζω λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ολοκληρωθεί το ολονομικό πλαίσιο. Θα επεκταθεί και στον έξω κόσμο τρόπον Α, θα συμπληρώσει τη σύμβαση του Λουγκάνο, τη σύμβαση που έχουμε με την Ισλανδία και την σύμβαση για την επιλογή δικαιοδοσίας η οποία κυρώθηκε επίσης πέρσι. Από την πλευρά μας λοιπόν συμμετέχουμε πλήρως στην όλη αυτή προσπάθεια και είμαστε βέβαιοι ότι θα ευοδοθεί τους επόμενους μήνες. και θα γίνει ένα πολύ σημαντικό μέρος της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σκέλος των δικαστικών θεμάτων και της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία μου. Συνάδελφοι, θέλετε το λόγο για το θέμα αυτό που μας παρουσίασαν οι δύο ε, εξαίρετες προκεκριμένες μας. Όχι, από ό,τι φαίνεται μας κατέκλυσε η το υπέροχό σα έργο. Γι' αυτό λοιπόν θα προχωρήσουμε στη συζήτησή μα και θα συνεχίσουμε με την ημέρα διάταξη. Επόμενο σημείο, μια έκθεση ε, που θα μα παρουσιάσει η κυρία Μπιόρκ εφόσον απουσιάζει ο κ. Μαστάλικα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχά θα μιλήσω αγγλικά. Οι σημειώσει που έχω είναι στα αγγλικά και θέλω να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου του κ. Μαστάλικα που δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα λόγω ζητημάτων υγείας, μου ζήτησε να σας παρουσιάσω απλώς τις βασικές του απόψεις για το όλο θέμα, για την εφαρμογή της οδηγίας 2004 του για την ε, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών. Εδώ η ισότητα των φύλων πρέπει να ε, ισχύει και σε άλλους τομείς της ζωής πέραν από τον εργασιακό χώρο, ωστόσο δεν έχει πλήρως ε, επιτευχθεί ο στόχος της οδηγίας. Κατά την άποψη του κ. Μαστάλκα, ε, θα πρέπει να περιοριστεί η έκθεσή του στι νομικέ πτυχέ του όλου θέματο. Ε, στέκεται στη νομική βάση του θέματο και σκοπεύει να υποβάλει παρατηρήσει για την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Δικαίου για την ίσιμη μεταχείριση των φύλων με σχετικές δικαστικέ αποφάσει του ΔΕΚ. Ιδίω αυτήν τη 30η Ιανουαρίου 2013 με την περίπτωση Τέστασα και την διατήρηση των βασικών αρχών στην περίπτωση των ασφαλιστικών κανόνων. Ο κανόνας UNISEX θα πρέπει να εφαρμόζεται στην περίπτωση των ασφαλιστικών απολαβών και αποζημιώσεων. Αυτό το θέμα το εξέτασαν και οι Επιτροπές ΛΥΜΠΕ και ΘΑΜ και κρίθηκε έκθεση τον Δεκέμβριο, γι' αυτό ο... θα εγκριθεί μέλλον τον Δεκέμβριο. Γι' αυτό ο κύριο Μαστάλκα για τη δική μα επιτροπή προτείνει το εξή χρονοδιάγραμμα. Δεν συνεδριάζουμε το Δεκέμβριο, θα πρέπει λοιπόν να την εγκρίνουμε τον Νοέμβριο. Το σχέδιο θα πρέπει να είναι έτοιμο για τις 7-8 Νοεμβρίου και η ψηφοφορία να λάβει χώρα στην Επιτροπή Νομικών Αποθέσεων στις 28-29 Νοεμβρίου. Με αυτά λοιπόν και με αυτά θα κλείσω εδώ, θα κρατήσω σημειώσεις, θα τις παραπέμψω στον κύριο Μαστάλικα και α, αν υπομονώ να ακούσω τις απόψεις των σχεδόν Η Επιτροπή θέλει το λόγο. Δεν ζητά το λόγο. Α, με συγχωρείτε κυρία μου. Ευχαριστώ. Ναι. Μια πολύ σύντομη παρατήρηση να τονίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν λάβει μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας αυτής στην χώρια νομοθεσία τους και για να προσαρμόσουν τις διαδικασίες τους καθώς και τους φορείς τους για τη σωστή της υλοποίηση. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το πώς προχωρούν όλα αυτά και να στηρίζουμε τα κράτη-μέλη προκειμένου να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο πλήρες δυναμικό της την οδηγία και να υπάρχει πραγματική ισότητα των φύλων ανά την Ευρώπη. Σε αυτή τη φάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί απαραίτητο να προτείνει τροπολογίες ή τροποποίηση στην οδηγία, αλλά θα δώσει προτεραιότητα στο να αντιμετωπίσει τα κενά και τις ελλείψεις στην μεταφορά της οδηγία, τα ενδεχόμενα σφάλματα, κυρίως ό,τι αφορά το πεδίο των εξαιρέσεων που προβλέπονται για την ε, εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Έχουμε εντατικούς διαλόγους, εντατικό διάλογο με αρκετά κράτη-μέλη για να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρχει σωστή υλοποίηση της οδηγίας. Η ισότητα των φύλων από την Ευρώπη και η σωστή υλοποίηση αυτή τη οδηγία σε όλα τα κράτη-μέλη είναι ένα θέμα που πραγματικά το έχουμε πάρει πολύ σοβαρά υπόψη και θα λάβουμε το ίδιο υπόψη και τι μέρημνε στο Ευρωκοινοβουλίου για να βελτιωθεί η κατάσταση τη ε, ισότητα των φύλων στην Ευρώπη. Επίση, Εξετάζουμε τις διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις για να καλυφθούν κάποια τα ζητήματα που θίγει η έκθεση με μια δυνατότητα ε, την μελέτη, να εκπονηθεί μελέτη για να μελετήσει τα θέματα αυτά, κάτι που έχει ήδη αναφερθεί και στις συζητήσεις σας στο Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν παρεμβάσεις. Ε, δεν βλέπω. Οπότε σας ευχαριστώ. Και θα σας δώσω το λόγο κυρία βιόρκα για το επόμενο θέμα. Ευχαριστώ. Και πάλι. Ήταν ευπρόσδεκτη η απόφαση να συμβληθούμε στην Σύμβαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση τη βία κατά των γενικών και τη ενδοοικογενειακή βία, την λεγόμενη Σύμβαση της ε, Ισταμπούλ, της Κωνσταντινούπολη, ε, και πάλι συγκεκριτής είναι ο κ. Μαστάλκα. Ε, εδώ και πάλι έχουμε κοινή έκθεση κοινέ αρμοδιότητες των Επιτροπών ΛΥΜΠΕ και ΘΑΜ. Έχουν ε, συμφωνήσει λοιπόν βάσει του άρθρου 55 δύο επιτροπές να ζητήσουν και την γνωμοδότηση τη δική μα επιτροπή. Εδώ στα χέρια μου έχω το χρονοδιάγραμμα για τη εργασίες των Επιτροπών ΦΑΜ και ΛΥΜΠΕ. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την έκθεση αυτή θα γίνει τον Ιούνιο του 2017 και η ψηφοφορία στις Επιτροπές ΛΥΜΠΕ και ΦΑΜ τον Μάιο του 2017. Οπότε η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων έχει αρκετό χρόνο μπροστά τη για να ετοιμάσει την γνωμοδότησή τη και ο κύριος Μαστάλκα θα ξεκινήσει τη σύνταξη και θα συνεισφέρει τις απόψεις του για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Αυτά προς στιγμή από μένα. Δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα ακόμη και δεν, έχουμε και να συμφωνή, δεν υπάρχει λόγος να συμφωνήσουμε για χρονοδιάγραμμα σήμερα. Ευχαριστώ κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω εκ μέρους της κυρίας Γκούτελαντ που δεν μπορεί να έρθει σήμερα οπότε απλώς θα διαβάσω την δική της παρέμβαση. Προσφάτως ε, ενημέρωσα για αυτά το... Προσφάτως ε, απέκτησα παιδί Κάτι που με δυσκολεύει στο να παραστώ σήμερα στις συζητήσεις ε, για το τόσο σημαντικό αυτό θέμα στην Επιτροπή Νίκολικοθέσεων με τι κοινέ εργασίε ΦΑΜ και ΛΥΜΠΕ. Ω και όδη από του σοσιαλιστέ και δημοκράτε το θέμα αυτό, θέλω να μοιραστώ μαζί σα όμω κάποιε σκέψει. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κυρώσει την ε, σύμβαση τη Ισταμπούλ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που υποβλήθηκε το Μάρτιο του 2016 βεβαίω είναι ένα σημαντικό βήμα για να προχωρήσουμε στα, στη λήψη των σωστών μέτρων όπω προτείνει η σύμβαση τη Ισταμπούλ για να καταπολεμήσουμε την ε, βία και τη διακριτή μεταχείριση βάσει των φύλων. Πρέπει να αναλάβουμε αποφασιστική δράση βάσει των αριθμητικών στοιχείων τη Επιτροπή. Μια στι τρει γυναίκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπάρξει θύμα σωματική ή σεξουαλική βία. Συνολικά 55% των γυναικών έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση και μια στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία από κάποιον ενήλικο κατά την παιδική τη ηλικία. Για να μην ε, αναφέρουμε τι υποθέσει που δεν έχουν καν καταγραφεί, εφόσον πολλέ φορέ τα θύματα όταν καν τα ε, λένε αυτά, τα καταγγέλνουν στην αστυνομία. Χρειάζεται εδώ κατεπίγουσα δράση από τα κράτη-μέλη και λήψη μέτρων, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα ανισότητα. Ε, η σύμβαση της Ισταμπούλ προτείνει μέτρα προς την πρόσβαση σε χώρου προστατευμένου, την ε, νομική και αστυνομική προστασία. Όμω κάποια από αυτά δεν θα έχουν αποτέλεσμα σε κάποιο μέρο, μέρη τη Επίρου μα αν δεν κυρώσουν την ε, σύμβαση με τα κάτι μελη Οπότε εμεί, ω μέλη τη Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, θα πρέπει να αποστείλουμε ένα χειρόπολιτικό πολιτικό μήνυμα προ τι Επιτροπέ Λίμπε και ΘΑΜ, ε, υπογραμμίζοντα την έντον, την πραγματική ανάγκη για τα κάτι μέλη και ε, τους αρμόδιους φορείς να εγκρίνουν την σύμβαση. Κυρία ε, Ντελβό, μας φέρετε δύο ευχαριστήσεις ειδήσει. Πρώτα απ' όλα, ε, την ε, τόσο συνοπτική παρουσίαση της κυρίας Γκούτλαντ και μετά φαίνεται ότι σήμερα γεμίσαμε μωρά. Με τόσο μεγάλη ταχύτητα, ο κύριος Ντυρόν προηγουμένως μας ανακοίνωσε τη γέννηση του δικού του παιδιού και τώρα μαθαίνουμε ότι και η κυρία Γκούτελαντ από τη χώρα της ε, έχει γίνει μητέρα. Να τη συγχαρείτε και, να τη εκείνη εκ μέρου μας, σας παρακαλώ. Και να ρωτήσω ποιο θέλει να παρέμβει τώρα για το επί τη ουσία ζήτημα. Τα όσα μα είπε ο εισηγητή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να επισημάνει. Ούτε εσεί συνάδελφοι. Παρακαλώ κύριε, έχετε το λόγο. Ήθελα απλώ να σα επισημάνω για όσους ενδιαφέρονται ότι θα διοργανωθεί σεμινάριο τον Νοέμβριο για το θέμα αυτό στις 23 του μήνα ε, συγκεκριμένα με θέμα την σύμβαση της Ισταμπούλ με, υπό την αιγίδα της Επιτροπής μας, της Επιτροπής των Δικαιωμάτων των Γυναικών και επίσης μια μελέτη πρόκειται να δημοσιευτεί για τα θέματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενημερωθούν όλοι. Ε, προσκαλώ λοιπόν τα μέλη της ε, Επιτροπής να συμμετάσχουν στις εργασίες μας. Ευχαριστώ. Άλλες παρεμβάσεις. Ωραία. Ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Ο κύριος Πασκάλ Ντουιγόν έχει το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ επίσης που μας δώσατε, που ανακοινώσατε το καλό νέο για το νεογέννητο. Είδα ότι είστε Γάλλος, έτσι. Είπατε μελλοντικό φορολογούμενος. Ε, ελπίζω να μεγαλώσει και να έχει τη χαρά να μεγαλούσε μια Ευρώπη ενιαία, αλληλέγγυα, την οποία δεν θα χωρίζουν, δεν θα διαιρούν οι εθνικισμοί. Αυτή είναι η ελπίδα μου για αυτόν και όχι να είναι απλά φορολογούμενος. Φορολογούμενος θα είναι ούτως ή άλλως. Να, είναι, να μεγαλώσει ως Ευρωπαίος και να ζήσει σε ειρήνη και δημοκρατία. Αυτά τα προσπαθούμε να οικοδομήσουμε καθημερινά. Και βεβαίως να πληρώνει τους φόρους του. Θα τους πληρώνει ελπίζω. Αποκλείεται να μην πληρώσει, λέει ο πρόεδρο. Ναι, ναι, είμαι πεπισμένο, λέει ο κύριο Ντυρό. Λοιπόν, λίγο πιο σοβαρά τώρα. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση πρωτοβουλίας ε, της κυρίας Καμπεθών Ρουίθ για την πρόσβαση στα φάρμακα. Και βεβαίως εδώ ε, μιλάμε για την πρόσβαση στην υγεία, στα φάρμακα, μιλάμε για κάτι εξαιρετικά επίκαιρο και βεβαίω είναι κάτι που αφορά και τη δημοσιονομική ισορροπία, διότι το κόστος ε, της υγείας ε, ε, είναι σημαντικό για του προπολογισμού. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τον τρόπο να χρηματοδοτήσουμε την υγεία και ταυτόχρονα οι πιο ευπαθείς ομάδες να μην αποκλείονται από την ιατρική περίθαλψη. Είναι θεμελιώδης αρχή αυτή των δημοκρατιών μας. Λοιπόν, δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Έγινε μια πολύ καλή μελέτη το 2009 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας επέτρεψε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει αυτή η απόκληση μεταξύ της, των τιμών των φαρμάκων και της ανάγκης ε, περίθαλψης και αποζημίωσης ε, ε, που τα συνοδεύουν. Το σκέλος των επενδύσεων που αφορούν στην έρευνα είναι πιο χαμηλό από τα ποσά που διατίθενται στη διαφήμιση και στο μάρκετινγκ. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε ένα απίστευτο παράδοξο. Η χρηματοδότηση, η αλληλέγγυα, πάει κυρίως σε εκστρατείες επικοινωνίας. Περισσότερο από ό,τι στην έρευνα. Αυτό είναι πρόβλημα. Είναι γνωστό το πρόβλημα αυτό, αλλά πρέπει να το επαναλάβουμε. Επιπλέον, υπάρχει και αυτή η δυσκολία διότι αφενός έχουμε την τιμή των φαρμάκων για αυτούς που έχουν τα, ε, τα δικαιώματα των φαρμάκων αυτών και από την άλλη έχουμε τα ε, φάρμακα τα γενώσιμα τα οποία είναι υπεραπαραίτητα στις κοινωνίες μας. Χρειάζεται λοιπόν ισορροπία. Αφενός έχουμε το κόστος και τα δικαιώματα που έχουν πάνω στα φάρμακα αυτά όσο τα παράγουν και αφετέρου δεν πρέπει να έχουμε ε, δεύτερα, τρίτα ε, διπλώματα ευρεστεχνίας που να μην μας επιτρέπουν τελικά να παράγουμε γενώσιμα ε, ο αριθμός των ε, δικαστικών αντιπαραθέσεων για ζητήματα αυτά έχει αυξηθεί δραματικά και συνήθω αυτά μικρά ε, εργαστήρια των γενώσιμων κερδίζουν, αλλά οι υπόλοιποι, οι μεγάλοι, κερδίζουν χρόνο. Διότι για όλο αυτό το χρόνο μέχρι να εκδικαστεί απόφα η απόφαση, τα μεγάλα εργαστήρια συνεχίζουν να αυγατίζουν τα κέρδη τους και τα γενώσιμα δεν μπορούν να απτυχθούν. Λοιπόν, υπάρχει μια μικρή αφίσα και να μην ξέρει κανείς γαλλικά, το βλέπει αυτό. Το 2014 είχαμε ένα φάρμακο για την υπαρήτητα ΓΑΜΑ. Πρόκειται για μια καμπάνια των γιατρών του κόσμου, έτσι. Ε, γιατρούς του κόσμου τους ξέρουμε όλοι. Ένα πολύ αποτελεσματικό φάρμακο λοιπόν για την υπαρήτητα Γ το οποίο πωλείται εντό εισαγωγικών, διότι υπήρξε διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Υγεία τη Γαλλία και με την κάθε χώρα, 41.000 ευρώ πωλείται το φάρμακο αυτό στη Γαλλία. Δεν μπορούμε να, να περιθάλψουμε όσους έχουν υπάρξει γάμα έτσι, οπότε υπάρχει επιλογή. Μόλις 1% των Γάλλων μπορούν να πάθουν υπαρτίδα γάμα, έτσι. Αυτό λέει η Αφίσα. Ε, λίγο προκλητικό ε, αυτό που λέει, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Θα πρέπει να επιλέξουμε ποιος θα λαμβάνει φάρμακο και ποιος όχι. Το κόστος του φάρμακου είναι 89 ευρώ. Το κόστος της, το κόστος της περίθαλψης. Αλλά είναι 41.000 το φάρμακο. Τέτοιου ζητήματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν. Και τελειώνοντας, Πρόεδρε, συγγνώμη αν μακρηγόρησα, αλλά το θέμα είναι σημαντικό. Προσπαθούμε στη γνωμοδότηση αυτή να πούμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα κείμενα που έχουμε στη διάθεσή μας, όλα τα νομοθετήματα, έτσι ώστε να έχουμε υποχρεωτικές άδειες ιδιαίτερα για την υπαρήτηδα Γ, είναι αυτό ακριβώς που επιτρέπει στα κράτος μέλος να επιβάλλει την χρήση αποζημιώνοντας βέβαια, αλλά πρέπει το εργαστήριο είναι υποχρεωμένο να διαθέσει το φάρμακο αυτό με αντίτιμο μία ε, ε, αποζημίωση δίκαιη, όπως όταν γίνεται μια παλωτρίωση για να φτιαχτεί ένας δρόμος, ένα αεροδρόμιο. Το φάρμακα είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικά με ένα αυτοκινητόδρομο ή ένα αεροδρόμιο. Δεν χρειάζεται νομίζω να σας πείσω γι' αυτό. Και το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να πείσω την προσοχή της Επιτροπής σας, τα κριτήρια για το κατά πόσο ένα φάρμακο μπορεί ε, να ε, χαίρει ενός διπλώματος και το κατά πόσο γίνονται σεβαστά τα κριτήρια αυτά είναι είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Οι γιατροί του κόσμου το λένε αυτό, για το, ειδικά για το φάρμακο την υπαρτίδα Γ. Πρέπει να φροντίζουμε αυτά τα χαρακτηριστικά για το κατά πόσο ένα φάρμακο πρέπει να χέρει προστασία ε, γίνονται σεβαστά. Ευθύ εξ αρχή πρέπει να μπορεί να γίνει αυτό και όχι να, να παρεμβαίνουμε μετά εκ των υστέρων. Και το τρίτο που ήθελα να πω και που αναφέρω στη γνωμοδότηση, η χνηλασιμότητα, διαφάνεια των δεδομένων, να μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει όλα τα στοιχεία στη διάθεσή της, Όπως βλέπετε δεν έχει τίποτα επαναστατικό αυτή η γνωμοδότηση. Προσπαθούμε απλώς να επιφέρουμε εκ νέου μια ισορροπία, να εξορροπήσουμε λίγο τα πράγματα, διότι υπάρχει μια προσέγγιση όλο και πιο εμπορική και η υγεία, ιδιαίτερα των πιο φτωχών της Υπήρου μας, διακυβεύεται έτσι. Μάλιστα, αγαπητέ συνάδελφοι, μπορείτε με μια φράση να μας επεξηγήσετε σε ό,τι φορά αυτά τα χαρακτηριστικά ε, κατά, πόσο ένα φάρμακο έχει, ε, πρέπει να χέρει ενός διπλώματος προστασίας, ευαισθητεχνίας ή όχι. Ναι, δεν ήθελα να μπω στις ε, λεπτομέρειες της μελέτης, αλλά φέρετε πάντως στη μελέτη που έκανε η Κομισιόν το 2009. Υπάρχει Καταρχήν ε, το κριτήριο του κατά πόσο ε, είναι ε, πρωτότυπη, πρωτότυπο αυτό το, το φάρμακο. Γι' αυτό κάνει αγωγή αυτή τη στιγμή για το φάρμακο την υπάτητα γάμα η οργάνωση γιατρή του κόσμου. Διότι το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη ουσία δεν ανήκει κανονικά στο εργαστήριο αυτό. Και δεν είχε γίνει έρευνα ούτε εφαρμοσμένη έρευνα, ούτε βασική έρευνα για την Πατρίδα γάμα. Πήρε δηλαδή ένα γνωστό ήδη, ε, μια γνωστή ουσία για να την εφαρμόσει την υπατήδα Γ. Έχω όλα τα στοιχεία στη διάθεσή μου και μπορώ να σας τα δείξω. Σε γενικές γραμμές πάντως αυτό που θέλουμε είναι τα κριτήρια που θα διέπουν ε, τα διπλώματα προστασία των φαρμάκων θα είναι, να είναι τα ίδια για όλου και να εφαρμόζονται. Διότι τις πρώτερες, τις τι δίκες τις κερδίζουν αυτοί που φτιάχνουν γενώσιμα. Τα κερδίζουν. Δηλαδή τα, τα συγκεκριμένα διπλώματα δεν ήταν έγκυρα. Ή εν ήταν πολύ περιοριστικά. Ή ενδεχομένω ε, δημοσίω. Ήταν δημόσια, λέει ο πρόεδρο. Ναι, βεβαίω. Διαπιστώνουμε ότι στι χώρε του Νότου ή στι αναπτυσσόμενε χώρε χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο να εδώ ας πούμε, για αυτό το φάρμακο, συγγνώμη δεν είναι μονή, αλλά ταιριάζει εδώ, η κυβέρνηση της Ινδίας έκανε αυτό που είπα πριν. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο έγινε μια παλωτρίωση. Δηλαδή, το κράτος, το κράτος μπόρεσε να προμηθευτεί το φάρμακο αυτό ε, σε λογικές τιμές με κάποια λογική αποσημείωση για το εργαστήριο. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη προσέγγιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλει κάποιο το λόγο, η κυρία Λί. Είναι σκιώδης η συγκέντρια, μάλιστα. Όπως ανέφερε ο συνάδελφος, σε σχέση με το αίτημα που είχε ε, εκτεθεί σε αυτό το σχέδιο, ζητείται να υπάρχει προστασία της ιδιωτικής ε, περιουσίας. Αλλά εδώ υπάρχει και η πτυχή των φαρμακευτικών προϊόντων. Και τώρα σε σχέση με την αύξηση των τελευταίων δεκαετιών, πράγμα το οποίο μπορεί να σημαίνει ένα περιορισμό σε σχέση με πρόσβαση σε φαρμακευτική αγωγή, καθώς επίσης και για τα γενώσιμα όσον αφορά για παράδειγμα καταχρηστική χρήση πολλές φορές ή κατάχρηση του συστήματος πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορά επίσης και αυτό κάτι πολύ σημαντικό και που μπορεί να καθυστερήσει την πρόσβαση των γενοσύμων στην αγορά. Και για αυτή την ε, τροπολογία που τον Οκτώβριο θα εξεταστεί, Εμεί θα καταθέσουμε αρκετέ τροπολογίες. Ευχαριστώ για το έργο του εισηγητή. Υπάρχουν ε, σημεία στα οποία μπορεί να υπάρχουν παρεκκλίνουσες απόψεις όσον αφορά τα δημόσια συμφέροντα και τα ιδιωτικά συμφέροντα για την διασφάλιση στην πρόσβαση. Υπάρχει όμως και το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και πρέπει να εξεταστεί και αυτό, διότι υπάρχει το θέμα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών και υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις, πράγμα το οποίο αφορά την, ιδιωτική, την πνευματική ιδιοκτησία. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η αηφορία των υγειονομικών συστημάτων όμως και είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό να υπάρχουν κίνητρα και το θέμα των ευρεσιτεχνιών είναι πάρα πολύ σημαντικό ώστε να μπορούν να έχουν τα ωφέλη για το έργο τους ε, οι δημιουργοί οι, όσοι έχουν ε, προβεί σε τέτοια ευρεσιτεχνία. Και ταυτόχρονα πρέπει να μπορούμε να προαγάγουμε και την έρευνα όσον αφορά τα φάρμακα. Και γι' αυτό πρέπει να προστατεύεται η πνευματική ιδιοκτησία. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν και θα πρέπει να συνεισφέρουμε καταθέτοντας τροπολογίες για τη βελτίωση του κειμένου για να υπάρξει ισορροπία. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, madame. Euh, madame Lee, pour la Commission européenne, s'il vous plaît. Ευχαριστώ, κυρία Λί, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι, όπως είπαν οι ευρωβουλευτές, Πρέπει να βρεθεί το σωστό σημείο ισορροπία στην Ευρώπη μεταξύ των κινήτρων που δίνονται για την έρευνα και την ανάπτυξη και την ε, ισότιμη πρόσβαση στα φάρμακα και τα βιώσιμα συστήματα υγεία. Δεν είναι εύκολο αυτό. Είναι συλλογική ευθύνη όλων μα, την οποία μοιραζόμαστε σε, σε, σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνηση, εθνικό, ευρωπαϊκό, τοπικό επίπεδο. Θα γνωρίζετε ότι στο Συμβούλιο Είχαμε το συμπέρασμα της 17ης Ιουνίου σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τα διπλώματα, τις πατέντε, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο για την καινοτομία. Ε, χρειαζόμαστε δηλαδή καινοτόμα φάρμακα, ε, διότι και ο πληθυσμό Ευρωπαϊκό γυράσκει, όμω οι αποφάσει πρέπει να παίρνονται με βάση συγκεκριμένα αυτά στοιχεία και προσπαθούμε να δώσουμε κίτα, να εξετάσουμε τα κίνητρα που δίνονται και να δούμε πώς αυτά βοηθούν στην καινοτομία χωρίς να παρεμποδίζουν την προσβασιμότητα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το φαρμακευτικό τομέα και την έκθεση του 2009 και τις σχετικέ εκθέσεις που ακολούθησαν σε ό,τι αφορά την επίλυση διαφορών για τις πατέντες, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά ε, το γηγείο ανταγωνισμού. Ε, πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση των στοιχείων της κάθε πατέντας πριν φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι εδώ υπάρχει παραβίαση του δικαίου ανταγωνισμού. Και σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα, η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο η αξιολόγηση της ασθένειας για να δούμε ε, κατά πόσο το ποσό που ζητείτε είναι το κατάλληλο. Πρόσφατα υπήρξε σχετική έγκριση στην αξιολόγηση αντικτύπου. Ε, εμείς θεωρούμε ότι ο μηχανισμός διαφάνειας θα επιτρέψει καλύτερη πρόσβαση στα φάρμακα και θα επιτρέψει να έχουμε μια, ένα πιο βιώσιμο σύστημα. Η Κομισιόν έχει πολύ περιορισμένες αρμοδιότητες στον τομέα αυτών, αλλά ζητούμε συνεργασία με τον κρατό μελών. Αναμένουμε το αποτέλεσμα αυτής της μόλι πρωτοβουλίας και υποστηρίζουμε ε, τους εισηγητές και τους ευρωβουλευτές που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Merci beaucoup, madame. Madame Regner la parole. Ευχαριστούμε, κυρία Ρέγνερ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο σκιώδης εισηγητής ε, Ενρίκο Γκαρπάρο δεν μπορεί να παραστεί. Θα προσπαθήσω να διαβιβάσω αυτά τα οποία προετοίμασε και τα οποία συμμερίζομαι. Η ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών, η ομάδα μας ε, ε, είναι ικανοποιημένη με την γνωμοδότηση που είναι καλή συνεισφορά και καλύπτει πολλές ε, προτεραιότητες όσον αφορά την πρόσβαση και διάθεση φαρμάκων. Και είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούν οι δεσμεύσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ιδιαίτερα από την έναρξη αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας υποστηρίζοντας μια ευρύτερη πρόσβαση σε φάρμακα. Η πρόσβαση στα φάρμακα δεν είναι απλά μια πολιτική που έχει συνταγματική αξία ως αρχές που καθορίζονται από τη συνθήκη και από την Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και φυσικά τα θέματα όσον αφορά τις ευρεσιτεχνίες ε, πρέπει να βοηθήσουν να είναι η έρευνα πιο ελκυστική. Αλλά πρέπει επίσης η καινοτομία να μπορεί να προαχθεί όσον αφορά τα φάρμακα και την μέρημνα, ιδιαίτερα ε, και σε κάποιους ε, σπανιότερους τομείς. Καταχρηστικές στρατηγικές όσον αφορά την παρακόλληση ε, της αγοράς πρέπει να αποφεύγεται. Ιδιαίτερα εμείς οι σοσιαλδημοκράτες δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο διαρκές πρασίνισμα, evergreening σε σχέση με μικρές τροποποιήσεις ε, υφιστάμενων προϊόντων ώστε να, παραταθούν, ή να παραταθεί η διάρκεια διαρκεια τεχνιών και να μπορέσουν να παράγονται. Ε, υπάρχει προτεραιότητα σε αυτό το τομέα και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει νέα προώθηση όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 89 ώστε να μπορέσει να έχει η αγορά τα φάρμακα αυτά στις ε, προσιτές τιμές και να κάνει μια προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να ενημερώνεται το κοινό και να μπορεί αυτό να καλύψει τις ανάγκες. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και εξ του κυρίου Γκασπάρα σας διαβίβασα ε, τις αφόψεις του. Ο κύριος Μαρίνιο παρακαλώ. Πιστεύω ότι αυτό, αυτή η περίπτωση είναι ένα υπόδειγμα, παραδειγματική περίπτωση. Στο μέτρο που μας οδηγεί να προβληματιστούμε για τις, τους κανόνες της αγοράς. Εγώ είμαι υπέρμαχος της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Όμως θα πρέπει να παρεμβαίνει το κράτος για να μπορεί να ρυθμίζει τις υπερβολές και ανεπάρκειες της αγοράς και στον τομέα ακριβώς των φαρμάκων εδώ και την πρόσβαση στα φάρμακα πραγματικά διακυβεύονται οι βασικοί κανόνες ε, της αγοράς. Μία επιχείρηση παράγει ένα προϊόν και το διαθέτει στην αγορά στην τιμή που επιθυμεί. Κάνουμε λοιπόν εδώ λόγο για φάρμακα και όχι για τέλη αεροδρομίων, για ταξίδια. Εδώ κάνουμε λόγο λοιπόν για περιπτώσεις καταχρηστικές, για κατάχρηση. Σε γενικούς όρους συμφωνώ με το, την προσέγγιση από πλευράς της έκθεσης του συναδέλφου Ντυρόν. Θέλω όμως να κρούσω κόδωνα κινδύνου ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξουν κάποιες προσαρμογές και κάποιες τροποποιήσεις θέλουμε πραγματικά ως άτομο με τις προόδους της ιατρικής και της επιστήμης στην ανακάλυψη φαρμάκων, στην επιστημονική, επιστημονική έρευνα κατά των ασθενειών. Και πραγματικά αναγνωρίζω αυτές τις προόδους και αναγνωρίζω ότι γίνεται από ιδιωτικά, ιδιωτικά εργαστήρια που κάνουν μεγάλες επενδύσεις. Αυτά επενδύονται και έχουμε αυτές τις πρόοδους. Τα κράτη ουσιαστικά δεν κάνουν καμιά επένδυση για αυτή την έρευνα και τις περισσότερες φορές κοινωνικοποιούν, είναι πιο έχουν την τάση να εθνικοποιούν ή να κοινωνικοποιούν αυτές τις έρευνες και αυτά τα αποτελέσματα φοβούμαι ότι μπορεί να υπάρξει κάποια υπερβολή κατάχρηση ή να υπάρχει κάποια υπερβολή που μπορεί να οδηγήσει εδώ σε προβλήματα για την έρευνα όσον αφορά αυτά τα πειραματικά εργαστήρια και την φαρμακευτική βιομηχανία. Οι επενδύσεις που κάνουν είναι γιγάντιες σε σχέση με τις δημόσιες επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα. Παγκόσμια κιόλας αυτό. Και πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό το στοιχείο τη στιγμή ακριβώς που τίθεται το ερώτημα που θέτει αυτή η έκθεση. Το κράτος πρέπει να μπορεί να παρεμβαίνει, πιστεύω, ώστε να μετριάζονται οι υπερβολές της αγοράς σε μια κατάσταση μονοπωλιακών καταστάσεων, σε μια κατάσταση δεσπόζοντος ρόλου στην αγορά, χωρίς όμως να, να δημιουργείται δυσπιστία όσον αφορά την ίδια τη φαρμακευτική βιομηχανία που μπορεί να διακυβεύει ή να ε, υπονομεύει τις γιγάντιες ε, επενδύσεις που γίνονται στην ε, έρευνα και στην προσπάθεια ανακάλυψης νέων απαντήσεων για τις ασθένειες ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλες παρεμβάσεις του θέματος. Δεν σας είδα. Παρακαλώ. Ε κυρία Μπριζερόν, ε, ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Η πρόσβαση στα φάρμακα είναι πραγματικά ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι ένα δικαίωμα παρόμοιο με αυτό στη στέγαση και στην εργασία τα ε, αποτυχημένα, τα, η πρόσβαση επιτυχή φάρμακα, σε αποτελεσματικά φάρμακα δεν είναι απλή. Ε, είναι πολύ ακριβά και αντικείμενα μονοπωλίων πολλές φορές, το ίδιο και για την έρευνα. Ευχαριστώ και συγχαίρω τον συνάδελφο για την προσέγγιση του σε ό,τι αφορά την εξέταση του θέματος των διπλωμάτων που προστατεύουν τα φάρμακα και για τις εξηγήσεις που μας έδωσε. Είναι σαφές ότι οι ορφανές ασθένειες, και το αναφέρω γιατί το έχω ζήσει προσωπικά, χρειάζονται έρευνε ιδιαίτερα δαπερνηρέ ε, για την ε, φαρμακευτική βιομηχανία. Και η φαρμακοβιομηχανία, ε, ό,τι εταιρεία και να είναι, αυτό που αποσκοπεί να έχει είναι το οικονομικό κέρδο. Είναι λίγοι οι καταναλωτέ αυτών των προϊόντων που πραγματικά αφορούν πολύ λίγους ανθρώπους, ώστε να μην είναι επικερδές, επικερδίσει όλη αυτή η έρευνα και προσπάθεια για τις φαρμακοβιομηχανίες. Και πολλέ φορέ τα φάρμακα αυτά δεν διατίθενται στι χώρε που τα χρειάζονται ή δεν επιστρέφονται τα χρήματα από το κόστο και πολλέ φορέ οι ασθενεί που πάσχουν από τι ορφανέ ασθένειε αναγκάζονται να προμηθεύονται αλλού. Είναι ε, επίση λίγε εγγυήσει ότι τα φάρμακα που υπάρχουν είναι πολύ αποτελεσματικά και πραγματικά χρήσιμα. Υπάρχει λοιπόν απόλυτη ανισότητα στην ε, πρόσβαση στα φάρμακα ω προ το αν είμαστε βέβαιοι ότι αντιμετωπίζουν μια συγκεκριμένη ασθένεια και να είναι ασφαλή. Κάτι άλλο που πάντοτε με ευνηδίαζε είναι η γενοδορία με την οποία τα φάρμακα ανακούφιση ε, συνταγογραφούνται πολύ εύκολα, είναι πολύ φτηνά και σε πολύ, κατά πολύ μεγάλο μέρο ε, επιστρέφονται και καλύπτονται από το σύστημα κοινωνική ε, πρόνοια. Μιλάω για τι παρακεταμόλε και τα ευουπροφέν. Ε, επειδή γνωρίζω και έχω ήδη φροντίσει ηλικιωμένα άτομα που έχουν χάσει ζωή τους, έχουν ε, φύγει πλέον από κοντά μας, ε, εκατοντάδες ε, κουτιά ντόλι κατανέλωσαν, είναι το δημόσιο τομέα φάρμακα αυτά, καλύπτονται, ε, όμως τα εργαστήρια αλλάζουν ένα μικρό γράμμα από τον τίτλο, το όνομα του φαρμάκου, με παρακεταμόλη κάποια άλλη αρωματική ουσία για να τα πουλήσουν αλλιώς με νέο δίπλωμα. Τα φάρμακα αυτά είναι συνήθως αναποτελεσματικότητα με ένα πολύ μικρό βαθμό ανακούφισης, αλλά αυτό το χρήμα που επιστρέφεται από το δημόσιο ταμείο για την ανακούφιση των ασθενών θα μπορούσε να αξιοποιείται για άλλους σκοπούς, όπως για τη στήριξη της έρευνας. Εκεί που χρειάζεται. Ε, είναι μια άλλη οπτική γωνία, αλλά νομίζω ότι είναι μια οπτική γωνία που θα ήταν χρήσιμη να την υιοθετήσουμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία μου. Άλλε παρεμβάσει. Από ό,τι φαίνεται όχι. Οπότε ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 29 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι και ε, αν θέλετε κύριε Ντυρό για το συμπέρασμα. Πολύ γρήγορα να ευχαριστήσω τους εξαιρετικούς μου συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους ε, που ήταν απεικοδομητικότατες. Απλώς δύο λόγια. Προφανώ, νομίζω το είχα πει ευθύ εξ αρχή και το επαναλαμβάνω, πρέπει να βρεθεί το σημείο ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων ιδιοκτησία και τη ανάγκη των εργαστηρίων ε, να αναπτύξουν φάρμακα που θα του επιτρέψουν να έχουν και οικονομικό κέρδο. Βέβαια, είναι επένδυση. Πρέπει να βρεθεί όμω το σωστό σημείο ισορροπία μεταξύ αυτού και του δικαιώματο στην υγεία. Ένα δικαίωμα που πρέπει να το προστατεύσουμε, ένα δικαίωμα για του πλέον μειονεκτούντε, για τι ε, σοβαρέ ασθένειε, για τι εμφανέ ασθένειε Ξέρουμε ότι πρέπει απλώς να βρεθεί το σωστό σημείο ισορροπίας. Η Βάλος ε, και εδώ μάλλον έχουμε έναν ιδιαίτερο ρόλο ως ε, συνομοθέτες, διότι η ιατρική έχει κάποιε ιδιαιτερότητε. Μιλάμε για τη μοναδικότητα ενός φαρμάκου, μιλάμε για φιλελεύθερο εμπόριο, αλλά στην Ευρώπη πρέπει να ε, δούμε αν η προσφορά και η ζήτηση μπορούν να εξορροπηθούν στην ίδια αγορά. Δηλαδή, ο γιατρό συνταγογραφεί, αλλά το κράτος δεν επιστρέφει τα χρήματα. Το εργαστήριο διαπραγματεύεται την τιμή του φαρμάκου με το κράτο και συζητώντα με, τον, με του γιατρού, τον ιατρικό κλάδο. Ο καταναλωτής όμως τελικά δεν ξέρει ποιον, τι πληρώνει σε ποιον. Ε, και ποια είναι η δική του η συμμετοχή. Είναι λοιπόν μια αγορά αυτών των φαρμάκων ε, που έχει σοβαρέ ελλείψει ισορροπία και εκεί πρέπει να παρέμβουμε, διότι δεν αρκούν οι ε, κανόνε ανταγωνισμού που ισχύουν κατά τα άλλα στην σημαντική παραδοσιακή αγορά. Αυτά νομίζω τα εξήγησαν και κάποιοι συνάδελφοι και για να απαντήσω στην παρατήρηση σε σχέση με το δικαίωμα μάλλον με το δίκαιο και του κανόνε που μπορεί να ισχύουν για, τον, για την ιδιοκτησία. Είμαι υπέρ του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών, όμω εδώ ε, υπάρχουν κάποιε ε, καταχρήσει και κάποια ιδίω ω προ την ε, προστασία κάποιων διπλωμάτων που δεν έχουν κανένα λόγο να θεωρηθούν ω τέτοια. Σα ευχαριστώ. Οπότε με την άδειά σα να περάσουμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διαταξή και πάλι μια έκθεση του κ. Ντυρό. Μια έκθεση που αφορά τα κριτήρια Ε, στην δήλωση συμφερόντων των Ευρωπαίων Επιτρόπων. Κύριε Τυρό. Ευχαριστώ Πρόεδρε κατά χρώμα του βέβαια, αλλά μετά θα σοπάσω, σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, έχουμε ξαναμιλήσει για το θέμα αυτό, δεν θα επανέλθουμε λεπτομερώς συνεπώς. Ε, ήθελα σε μια πρώτη φάση να πω, όταν είχα παρουσιάσει την γνωμοδότησή μου, έπρεπε ακόμα να περιμένουμε τις τροπολογίες, έτσι. Πρέπει να πω καταρχήν σε μια, μια πρώτη φάση ότι το σύνολο των τροπολογιών που έλαβα, ή αυτό σχεδόν το σύνολο, είναι εξαιρετικά σημαντικές τροπολογίες, διευκρινίζουν κάποια πράγματα, συμπληρώνουν, όχι μόνο ε, δεν αλλάζουν τη γνωμοδότηση προς το χειρότερο, δεν την επηρεάζουν αρνητικά, την βελτιώνουν και την ενισχύουν. Και αναφέρομαι στη δική σας τροπολογία, Πρόεδρε, για τον ορισμό του τι μπορεί να αποτελεί ε, σύγκρουση συμφερόντων ε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει να διευκρινίσει κάποια πράγματα. Ήθελα να πω ότι πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Το σύνολο των γνωμοδοτήσεων των τροπολογιών μάλλον έρχονται να βελτιώσουν το κείμενο. Ε, βεβαίως θα γίνουν κάποιες συζητήσεις με τους κοιόδους, με διότι κάποιες τροπολογίες ε, ενδεχομένως ε, να παρεμποδίζουν τη δυναμική που θέλουμε να δημιουργήσουμε εδώ, δηλαδή την, όσο γίνεται πιο πολεσματική καταπολέμηση των, ε, της σύγκρουση συμφερόντων, των διαπλεκόμενων συμφερόντων στο εσωτερικό της Ένωσης. Ε, πρόεδρε, δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα παράδειγμα εξαιρετικά δυσάρεστο σύγκρουση συμφερόντων, όπου διαπιστώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας, ε, της θητείας της ενός επίτροπος, μια επίτροπος που ε, αγοράζει μετοχές, ε, τις βάζει σε ένα φορολογικό παράδεισο χωρίς να τα δηλώνει πουθενά αυτά και θεωρώντας ότι δεν χρειάζεται να το κάνει. Επειδή όλα αυτά τελικά δεν είναι και τόσο σημαντικά. Είναι σημαντικά όμως. Είναι πολύ σημαντικά να το γνωρίζουμε. Αν τελικά δεν είναι σημαντικά, τότε δηλώστε τα. Γιατί τότε δεν δημιουργούμε πρόβλημα σε κανέναν. Λοιπόν, ας φροντίσουμε αυτή η εικόνα μιας Ευρώπης που έχει υποταχθεί υπερβολικά ε, στα ιδιωτικά συμφέροντα και όχι τόσο στο δημόσιο ε, δεν θα επικρατήσει αυτή η εικόνα, δεν θέλω να επικρατήσει οπότε θα τα ξαναζητήσουμε όλα αυτά στα πλαίσια μιας συνάντησης μεταξύ σκιώδων εισηγητών. Θέλει κάποιος το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Ράιτνερ. Ευχαριστώ και μπορώ και να τα πω αρκετά γρήγορα. Προσπαθούμε από την πείρα μας να καταλήξουμε στα σωστά συμπεράσματα από την πείρα που έχουμε συλλέξει σε σχέση με τις ακροάσεις επιτρόπων. Και θα έλεγα ότι όλη αυτή η έκθεση θα πρέπει να βοηθήσει ώστε να επιτελέσουμε το έργο μας ως Ευρωβουλευτές και να μπορέσουμε να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων, όχι μόνο τυπικά και με κάποια τυπικότητα να μπορέσουμε να δράσουμε. Αλλά να, είμαστε, να έχουμε ένα ευρύ πλαίσιο ε, χειρισμών και ελιγμών που θα δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας αρμοδιότητες και γι' αυτό με τροπολογίες πρέπει αυτό το στόχο να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Κύριος Χρυσόγονος παρακαλώ. Λοιπόν θα συμφωνούσα καταρχήν πρέπει να πω με τις απόψεις του εισηγητού και με την κυρία Ρέγνερ βέβαια. Είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια και έχω την εντύπωση ότι δεν είμαστε ικανοί, δεν είχαμε την προθυμία να πάμε όσο μακριά όσο έπρεπε να προχωρήσουμε στην τελευταία εξέταση των δηλώσεων των συμφερόντων των επιτρόπων και ιδιαίτερα όσον αφορά τη δήλωση συμφερόντων του Επιτρόπου για τα ενεργειακά θέματα. Αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να κάνει σωστά τη δουλειά που έπρεπε να κάνει, που πιστεύω και θεωρώ θα έπρεπε να κάνει, εξετάζοντας τα διαπιστευτήρια ε, των υποψηφίων. Οι γενικές κατευθυντηρίες γραμμές πρέπει να τίνουν προς μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο ενδελεχή εξέταση των δηλώσεων των επιτρόπων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό και πιστεύω ότι όλοι το παραδέχονται και το ομολογούν. Και είχαμε και τις ειδήσει ε, ε, της Bahama Leaks, ε, τις διαρροές από τις Μπαχάμες που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα και που όλα αυτά δείχνουν ότι είναι ένα πάρα πολύ επικαιρό θέμα αυτό. Όμως δεν βλέπω να διαγράφεται κάποια λύση, να διαφαίνεται κάποια λύση ως Ευρωβουλή θα πρέπει να θέτουμε ερωτήματα. Δεν μας αρέσει η κατάσταση ως έχει και για να την αλλάξουμε δεν ξέρω ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Έχουμε τρία επίπεδα. Υποβάλλονται συστάσεις για υποψήφιους επιτρόπους από τα κράτη-μέλη για αυτούς τους υποψηφίους. Διαρωτώ με, τα κράτη-μέλη που το κράτος μέλος που είχε συστήσει την Επίτροπο Κρούς. Ε, την περίπτωση αυτή την κάλυψε ικανοποιητικά. Δεν έχουμε μέσα και εργαλεία στα, στη διάθεσή μας και πολλές φορές ε, δεν υπάρχει και ιδιαίτερη τάση. Πώς μπορούμε να ασκήσουμε πίεση λοιπόν σε ένα κράτος. Πώς θα μπορούσαμε να δράσουμε ώστε να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχουν επαρκή στοιχεία για ενημέρωση και πληροφόρηση ώστε να μας, δίνει τη να μας δίνουν τη δυνατότητα μιας σε βάθος ανάλυσης. Ωστόσο όλοι συμφωνούμε σε αυτήν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή ότι δεν θέλουμε να είμαστε κατήγοροι ή εισαγγελείς και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από πλευράς εισηγητού. Φυσικά αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο έργο, εγχείρημα για τον Πασκάλ Ντουιρόν αυτό. Ωστόσο, θα ήθελα να τον ναι. ρωτήσω, να του ζητήσω σχετικά με αυτό, να λάβει υπόψη την πίεση που υφίσταται και που πρέπει να ασκηθεί στην Επιτροπή και στα κράτη-μέλη. Ο κύριος Μαρίνιο Πίν. Ε, ε, ε, Βλέπω ότι υπάρχουν δύο επίπεδα εδώ. Το ένα είναι στην πραγματική υλοποίηση των αρμοδιοτήτων αυτής της Κοινοβουλευτική Επιτροπής για την τον προηγούμενο έλεγχο όσον αφορά στοιχεία και ποσά που αφορούν τους Επιτρόπους Και συμφωνώ απόλυτα 100% με τον συνάδελφο Χρυσόγωνο. Δεν υλοποίησε η Επιτροπή σε σχέση με τον Επίτροπο που ανέφερε το έργο δεν είναι ένα εξειδικευμένο νομικό έργο η Επιτροπή, είναι ένα πολιτικό όργανο. Θα έπρεπε όμως να δημιουργηθούν μηχανισμοί αποτρεπτικοί τέτοιων πρακτικών να αποκρύπτονται τα συμφέροντα των Επιτρόπων αποστεριόρι ώστε να, υπάρχουν, να υπάρχει δυνατότητα επιβολής κυρώσεων που θα οδηγεί στο να μην ψεύδονται τα άτομα όπως ανακαλύφθηκε ότι εψεύστη μια πρώην επίτροπος σε σχέση με τα όσα είχε δηλώσει ή είχε ψευστεί, είχε ε, διαδώσει ψεύδι όσον αφορά τα συμφέροντά της σε υπεράκτιες εταιρείε. Πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις, πρόστιμα, αφαίρεση, στέρηση συντάξεων και προνομίων μια και υπήρξαν ψεύδι εδώ και έπρεπε να είχε αυτό το θέμα διευθετηθεί προηγούμενα. Γι' αυτό λοιπόν το να αφήνουμε τα πράγματα χωρίς να υπάρχει κανένα αποτελεσματικό μέτρο για κυρώσεις, για κύρωση, ε, αυτό θα μας δίνει απλά και μόνο θα ε, παρατείνει εσαΐ δηλώσεις και συζητήσεις χωρίς οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις, πρόστιμα για τα άτομα που δεν υλοποιούν τις υποχρεώσεις τους και αποκρύπτουν συμφέροντα και ψεύδονται όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά. Ευχαριστώ συνάδελφε. Άλλε παρεμβάσει όχι προ στιγμή. Ε, εάν με επιτρέπετε μια μικρή προσωπική παρατήρηση, θα μιλήσω όλε και καθόμουν εκεί. Κάντε ότι δεν το είδατε. Ξέρετε ότι είμαι πρώην δημοσιογράφος και ήμουν και αρχισυντάκτης και ήμουν και σε κανάλι, ιδιωτικό και κρατικό. Το κείμενο αυτό ε, πραγματικά αντικατοπτρίζει με τρόπο πολύ δυσάρεστο αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή, εδώ φαίνεται να επιτρέπουμε να ε, κυκλοφορούν πληροφορίες τις οποίες δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε. Πολλές από αυτές είναι και αναλυθείς. Δεν θυμάμαι να είχα να εξετάσω ψευδείς πληροφορίες από την άποψη της αλήθειας του ψεύδους, όμως είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά τουλάχιστον που ε, έχω πληροφορίες στα χέρια μου οι οποίες δεν είναι σαφώς πλήρεις και για τις οποίες πρέπει να εκφράσουμε μια έγκριση και να πούμε ότι μας ικανοποιούν υποψηφιότητε των Ευρωπαίων Επιτρόπων. Θα έλεγα ότι τα θεσμικά όργανα ε, δεν ε, δείχνουν καλή πίστη απέναντί μας, διότι δεν θα έπρεπε να εκβιαζόμαστε για κάτι για το οποίο δεν έχουμε πλήρη πληροφόρηση. Αυτό ισχύει ε, για τον Επίτροπο Αυτό ισχύει και για τον ε, έναν επίτροπο, αλλά και για την περίπτωση που, αναλάβατε, που αναφέρατε και όλα αυτά που συζητήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και να σα πω μια επιστολή που δεν δημοσιεύτηκε. Ότι το καλοκαίρι απέστειλα επιστολή στον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κώδικα συμπεριφορά. Ε, είναι το προήμιο, ένα παράρτημα μάλλον, δεν είναι το προήμιο. Ε, του ζήτησα ο κώδικα συμπεριφορά των πρώην επιτρόπων να αλλάξει, να τροποποιηθεί δεν είναι δυνατόν σε 18 μήνες να ανοίγουν τα σχήρα του οι επίτροποι και να λένε εντάξει είμαι πλέον ε, καθαρός και ξάστερος και αγνός άσπυλο. Θα πρέπει να ε, φροντίσουμε για την ουσία των νομοθετικών κειμένων που προωθούνται και προχωρούν, φεύγουν από το Κοινοβούλιο, πριν από λίγου μήνε, ξέρετε, ότι εγκρίναμε κείμενο το 2003-2004 κιόλα και βλέπουμε ότι κάποιε φορέ είναι τόσο μακροσκελής η κοιτάξει που οι επίτροποι πρέπει να προστατευτούν εφόσον έχουν εξετάσει τέτοια θέματα. Ακόμη και στο πλαίσιο μια ολοκλήρωση θητεία, μια πενταετία. Εντάξει, να αμυθούν, ε, γιατί όχι. Αλλά βλέπω ότι πραγματικά μα ε, έχουν φέρει σε θέση ε, δύσκολη που θα πρέπει να ε, μην εκβιαζόμαστε με τόσες ε, αλήθειες οι οποίες είναι ημιτελείς, το ίδιο και με ψεύδι, που ούτε αυτά μπορούν να ελεγχθούν. Να πω ότι όταν μιλάω για ψεύδι, εννοώ ότι μιλάω για ξεκάθαρα ψεύδι. Λένε ότι δεν έχουν πλέον κανένα συμφέρον πλέον πέραν αυτού που δηλώνεται. Ενώ στην πραγματικότητα υπήρχε συμφέρον. Σε αυτό λοιπόν το βαθμό, όταν κάποιο δηλώνει ότι τα μόνα του συμφέροντα είναι αυτά τα οποία έχουν δήλωθει, τα δεδηλωμένα και μετά ανακαλύπτω ότι υπήρχαν κι άλλα, αυτό αποτελεί ψεύδο. Ψεύδο κατάφορο και τελείω. Ε, ε, αντικειμενικό. Ε, στην περίπτωση που ανέφερε και η Ζέσκα και στα πλαίσια της δικής μας της ευθύνης, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει σοβαρότατη βλάβη ζημία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει μάλλον να προσεχθεί στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω με ποια μορφή δικαίου, αλλά δεν ξέρω και γιατί να το αφήσουμε έτσι. Σα ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση που μου δώσατε το δικαίωμα να πω την άποψή μου και να συνεισφέρω στη σύνταξη τη εκθεσή σα. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, κύριε ναι, ε, μόνο δύο κουβέντε, κύριε Πρόεδρε. Άλλη μια φορά θα ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου για τι συνεισφορέ του. Η συζήτηση πραγματικά δείχνει ότι είναι ένα θέμα που ε, είναι άκρο σημαντικό να στραφώ προς την κυρία Βριασκά, η οποία μου ευχήθηκε κουράγιο, θα τα πήγαινε και ίδια πολύ καλύτερα εάν μπορούσε ε, να συνεισφέρει στην προσπάθεια. Εάν προχωρήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι και καταλάβουμε ότι εδώ πρόκειται για ε, έναν σοβαρό πολιτικό σκοπό, θα πετύχουμε. Αλλά αν το δούμε ως πολιτικό παιχνίδι, μάλλον θα αποτύχουμε. Εδώ λοιπόν πρέπει να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπίας. Πρέπει να δούμε τι γίνεται μεταξύ του πώς λειτουργεί η πραγματικότητα, που δεν πηγαίνουν πάντα όλα υπέροχα και το τι συμβαίνει στον κόσμο τον ιδεατό τον κόσμο των ιδανικών. Πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε τον κόσμο του εφικτού. Δηλαδή από τη μια και την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να την καλέσουμε να σα απαντήσει. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κείμενα. Δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε δικαστηρίο μα, ούτε θέλουμε να κάνουμε ένα πραξικόπημα. Όμω υπάρχουν κείμενα τα οποία επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ε, ξαναδεί τον κώδικα συμπεριφορά των επιτρόπων. Σε αυτήν λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να απευθυνθούμε και να ζητήσουμε να ληφθούν υπόψη καθ' όλη τη διάρκεια τη θητεία λόγου χάρη τα οικογενειακά συμφέροντα ενδεχομένω ενό επιτρόπου. Δεν θα λειτουργήσουμε λοιπόν ω δικαστήριο, αλλά όπω άλλα κοινοβούλια ανά τον κόσμο, μπορούμε να ζητήσουμε να δοθούν απαντήσει για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, μια συγκεκριμένη υπόθεση και να μα δίδονται αληθεί πληροφορίε προτού περάσουμε στην επόμενη φάση. Αυτήν την ισορροπία νομίζω πρέπει να επιδιώξουμε και πραγματικά έχοντα ξεκάθαρα κατά νου ότι αυτά τα θέματα, αυτέ οι υποθέσει συγκρούσεων συμφερόντων που πολύ συχνά δημοσιεύονται στον τύπο το τελευταίο καιρό, πλήττουν την η καλή εικόνα τη Ευρώπη ούτω ή άλλω και νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι. Σα ευχαριστώ πολύ. Έγκριση τη έκθεση 13 Οκτωβρίου. να σας παρακαλέσω να τροποποιήσουμε και πάλι λιγάκι την ε, σειρά της ημέρας διαταξής, γιατί έχουν έρθει πολλοί συνάδελφοι ήδη για τις ψηφοφορίες και θέλουν να φύγουν μετά. Οπότε, αν με επιτρέπετε κύριε Καρύμ, μπορούμε να ε, συζητήσουμε την εκθεσή σας αμέσω μετά τις ψηφοφορίες. Πρόεδρε, έχω άφθονο χρόνο μπροστά μου, ε, όπως ξέρετε ειδικά αυτόν τον καιρό και η παράκλησή σας για μένα είναι διαταγή. Με, χαρά, με τα χαρά να μείνω. Πολύ ωραία. Οπότε ο κύριος Φάραντ σίγουρα θα δει και τα θετικά αυτή τη υπόθεση από τη δική του σκοπιά. Παρακαλώ ένα-δυο λεπτά ε, για να περάσουμε στις ψηφοφορίες, να βρουν όλες τις κάρτες τους, να καθίσουν. Παρακαλώ ελέγξτε αν έχετε μαζί τις κάρτες σας. Διακόπτουμε για δένα δίλεπτο. Συνάδελφοι, είστε έτοιμοι όλοι. Έχετε όλοι κάνει τη δοκιμή με τις κάρτες σας. Ωραία, ευχαριστώ. Πρώτη ψηφοφορία για την έκθεση του κυρίου Χρυσόγονου. Εάν θέλετε κύριε Χρυσόγονε να ασχοληθείτε. Ξεκινούμε με τη δική σας έκθεση. Ωραία, ευχαριστώ. Παράγραφος 1. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ευχαριστώ. Συμμεβαστική 6. Υπέρ. Κατά εποχές Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ευχαριστώ. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ευχαριστώ. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ευχαριστώ 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σας ευχαριστώ πολύ θα μπορούσαν οι διάφορες ε, γραμματείες, οι συνεργάτες να μην συζητούν ε, τόσο ψιθυριστά διότι ακούγονται στα μικρόφωνα και ενοχλούν. Θα σας παρακαλούσα να είστε σιωπηλοί. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 9. Συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Συμβαστική 10. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πέντε. Όχι. Πούντο. Α, ναι. Με συγχωρείτε. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα η σωστή σειρά. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ευχαριστώ, εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Υπέρ. Κατά. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η πληροφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμφωνούμε, δεν ξεχάσαμε κανένα, να λυθούμε σωστοί. Ναι, 18 και 4, σωστά, οπότε απορρίπτεται. 23, υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε στην έκθεση όπως τροποποιήθηκε. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία έρχεται. Πέρασε, ψήφισαν άπαντε. 20 υπέρ, 2 κατά, καμία εποχή. Ευχαριστώ, εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια στον συνάδελφο. Και τώρα περνάμε στην ψηφοφορία. της κυρίας Χάουταλα. Je vais essayer de comprendre ce que je n'ai Προσπαθώ να καταλάβω κάτι που δεν ε, κατανόησα. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο παρακαλώ. Avant le vote... Πριν την ψηφοφορία, κάποιος έχει ζητήσει το λόγο. Όχι, δεν θα δώσουμε το λόγο. Θα χαιρετήσουμε τον πρέσβη παρά την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κύριο Τουτσέσκι. Ήθελα πολύ να σας δω και διαζώσεις. Καλώς ήρθατε κύριε πρόεδρε. Κι επού; Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τόσο το χειρότερο για μένα. Έχει αστείο κατάλογο. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε πέρα τη ψηφοφορία. Αποτέλεσμα 19 υπέρ, 3 κατά, καμία εποχή. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε το σύνολο, όπω τροποποιήθηκε, του κυρίου Τσαμπάσκη. Αντιρρήσει. Ψηφίζουμε τα τρία τμήματα συνολικά ή το καθένα ξεχωριστά. On block, on block. Επειδή μου, έκανε, αρνητικά η κυρία Ρέγνερ, on block. Και με ονομαστική ψηφορία. Με γολ κολ. Άρχεται η ψηφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Ομοφωνία από τις λίγες. 22 υπέρ, καμία αρνητική ψήφους, καμία αποχή. Σας ευχαριστώ. Τελευταία ψηφοφορία. Νομική βάση. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να σχολιάσω, μην χάνουμε χρόνο. Και πάλι συστήνω αυτή τη νομική βάση. Ψηφίζουμε στην. Ε, περνάμε στην ψηφοφορία υπέρ. Κατά. Κατά. Α, να ένα. Αποχέ. Εγκρίνεται κανένα σχόλιο περί του εισηγητού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε αυτή την πρώτη σειρά ψήφων και τώρα θα ψηφίσουμε και κλεισμένο των θυρών για τις άρσεις ασυλίων. Περνούμε λοιπόν στη συνέχεια της συνεδρίασής μας. Και θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Καρίμ για το θέμα της επικορικότητας. Κύριε Καρύμ. Να ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά είμαι και πάλι συγγητής ε, σε αυτό το θέμα της ημερησίας διάταξη ε, για το, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα σε σχέση με το 2014. Σύντομα θα ήθελα να σκιαγραφίσω τις κυριότερες προτάσεις ε, στην πιο τελευταία μου αυτή έκθεση και θα περάσω με τα σημεία τα οποία... Συγγνώμη κύριε Καρύμ. Με συγχωρείτε να παρακαλέσω τους συναδέλφους που βρίσκονται ακόμη στην αίθουσα και τους επισκέπτε. Δεν είναι η πλατεία του Λουξεμβούργου εδώ και ο εισηγητής χρειάζεται την ησυχία του και οι διερμηνείς δεν έχουν αρκετή ηρεμία για να κάνουν σωστά τη δουλειά του. Παρακαλώ, χρειαζόμαστε ησυχία από την αίθουσα. Θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω διάφορα ευρήματα και προτάσεις που θεωρώ ότι ε, είναι ιδιαίτερα σκόπιμα. Πρώτα η επικουρικότητα και η έλεγχη μπορεί να θεωρηθούν ένα σημαντικό μέσο για να μειωθεί το δημοκρατικό έλλειμμα και να διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται όσο το δυνατόν κοντύτερα προσεγγίζοντας τους πολίτες σε σχέση με μια βήμα προς βήμα προσέγγιση που υιοθετήθηκε σε σχέση με το ευρωπαϊκό επίπεδο για μια ολόκληρη σειρά ετών. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο κάποια από τα εθνικά κοινοβούλια ανέφεραν ότι οι νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν ε, δικαιολογούν επαρκώς, δεν ε, καλύπτουν επαρκώς την αναλογικότητα και επικουρικότητα και υπάρχει εντύπωση ότι αυτή η έλεγχη είναι ανύπαρκτη ή δεν εφαρμόστηκαν καν καθόλου. Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία απορρέουν. τα εθνικά κοινοβούλια ζήτησαν μια <clears throat> 8 εβδομάδων περίοδο για τις αιτιολογημένες γνώμες και αυτό είναι κάτι σημαντικό επίσης. Όσον αφορά την Επιτροπή, όσον αφορά τη μελέτη επιπτώσεων, για τις ε, μελέτες που έχουν ε, συνταχθεί όσον αφορά το 2014 ανεπαρκής αναλύσεις αρχό, της αρχής της ε, επικουρικότητας και της αναλογικότητας έγιναν και υπάρχει γενικά εντύπωση ότι πολλά περισσότερα πρέπει να γίνουν για να εφαρμοστούν οι αναγκαίες ε, δοκιμασίες και έλεγχοι όχι απλά από εμάς αλλά και από τα αδελφά θεσμικά όργανα. Επίσης όσον αφορά την ε, εξέταση των συνθήκων και τον αριθμό των απαντήσεων που απαιτούνται από τα Εθνικά Κοινοβούλια για να ξεκινήσει η διαδικασία μιας κίτρινης κάρτας ή μιας πορτοκαλί κάρτας και για το συμπέρασμα αν μπορεί μια κόκκινη κάρτα να αρχίσει να λειτουργεί, αν ένας σημαντικός αριθμός εθνικών κοινοβουλίων εκφράσουν ανησυχίες ε, για το θέμα της επικουρικότητας, όλα αυτά δημιούργησαν, προκάλεσαν μια πολύ ε, θερμή πολιτική συζήτηση και υπάρχει μια ε, σταθερή στάση επ' αυτών ε, και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Για την ιδέα τώρα της πράσινης κάρτας ε, που θα μπορούσε να εξεταστεί δίνοντας στα Εθνικά Κοινοβούλια την ευκαιρία να εισαγάγουν νομοθεστικό έργο, να το απορρίψουν ή να το τροποποιήσουν και αυτό εξακολουθεί να βρίσκεται σε μεγάλο ε, βαθμό υποσυζήτηση. Θα με ενδιέφερε να ακούσω τις απόψεις των ε, συναδέλφων. Πολλές φορές γίνεται λόγος για την ε, αναλογικότητα και πρέπει εδώ να ληφθεί υπόψη και η αναλογικότητα και η επικουρικότητα και ζητούμε να υπάρξουν διευρυμένες ε, μελέτες επιπτώσεων ε, ε της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε, προτάσεις, σε προτάσεις που ε, δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά επιβαρυντικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αιτιολογημένες γνώμες θα πρέπει να εξετάζονται από τα Εθνικά Κοινοβούλια σχετικά και να δούμε τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ισχύουν, μήπως μη δεσμευτικέ ε, κατευθυντήρες γραμμές και προσανατολισμοί θα πρέπει να εκπονηθούν για να μπορούν να ακολουθηθούν τέτοιες, ε, ε, τέτοιοι προσανατολισμοί για την επικουρικότητα και αναλογικότητα. Όλα αυτά σε στενή διαβούλευση πάντα με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα είδατε από την παρουσίαση που έκανα απόψε συνάδελφοι ότι δεν προσπάθησα να παρουσιάσω τις δικές μου απόψεις όσον αφορά τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Πάντα ήταν η άποψή μου ότι σε πολλά επίπεδα πρέπει να διατεθεί, να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα ώστε να μπορούν ε, τα εθνικά κοινοβούλια σε σχέση με τους πολίτες ε, να ε, παρουσιάζουν το έργο και να μην αφαιρείται από αυτά το έργο και να διευρύνεται η δυνατότητα σε σχέση με την παρέμβαση και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ ως Βρετανός Ευρωβουλευτής μην έχοντας επιβάλει αυτή την ημερήσια διάταξη, η στάση μου πάντα ήταν ανοιχτή, αλλά τώρα πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο ανοιχτή σε σχέση με το παρελθόν για να διασφαλίσουμε ότι οι απόψεις των συναδέρφων που πραγματικά θα εργαστούν στο μέλλον θα πρέπει να ληφθούν υπόψη έγκαιρα και εύθετα. Ευχαριστώ. Merci beaucoup de... Σας ευχαριστώ πολύ για την τόσο ισόρροπη παρουσίαση και για αυτό που είπατε συμπερασματικά. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να χαιρετήσω την έκθεση του συνάδελφου Τσακαρίν που πάει προς σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την ε, προστασία των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Συμμερίζομαι και το έχω ξαναπεί τις ανησυχίες ε, σχετικά με τις ανεπαρκείς ή ανύπαρκτες ε, αιτιολογήσεις για το θέμα αυτό στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το ίδιο ισχύει και για την ανεπάρκεια των, των αναλύσεων αντικτύπου. Χαιρετίζω τι προτάσει σα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εισαγωγή μια κόκκινη κάρτα και μια πράσινη κάρτα, Θα ήθελα να προσθέσω ότι η προθεσμία για ένα εθνικό κοινοβούλιο για να ε, ε, δώσει αιτιολογημένη άποψη είναι πολύ μικρή και πρόκειται για μια διαδικασία που πρέπει να ισχύει για το σύνολο της νομοθετικής διαδικασίας ή τουλάχιστον να μπορεί να γίνει στα μέσα της διαδρομής και στο τέλος της διαδικασίας. Ε, Τώρα από εκεί πέρα εγώ είμαι ε, λίγο πιο εχμηρή από εσά. Πρέπει να γίνουμε πιο επιθετικοί απέναντι στην Κομισιόν που όταν ένα κράτος μέλος δεν σέβεται τις ε, υποχρεώσει του ε, αυτή το επισημαίνει. Τα προβλήματα όμως ισορεύονται χωρίς να υπάρξει καμία βελτίωση. Αυτή η αρχή της επικουρικότητας είναι ο φτωχό συγγενής. Αυτό το σύστημα είναι αμυγός αντιδημοκρατικό δεν έχω αυταπάτες. Η έκθεσή σας ε, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να ακολουθήσει μια τέτοια οδό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Και τώρα ο κύριος Βζιέσκα ή η κυρία Ντελβό. Πρώτα ίσως. Ο κύριος Βζιέσκα έχει στήσει το λόγο πριν. Όχι, δεν θέλει, δεν θέλει. Κύριε Βιέσκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. ή από πλευρά της ίσως θα, θα ακολουθηθεί η άποψη μου. Είναι ιδιαίτερη χαρά να συνεργαζόμαστε με τον κύριο Κάρη για την συνέπεια και συνεκτικότητα που χρειαζόμαστε. Αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα καθημερινά και όχι μόνο στο επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου και σε σχέση με το ευρωπαϊκό δίκαιο αλλά και σε σχέση με τις χώρες μας, τα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να επιληθούν αυτά τα προβλήματα και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να τεθεί σε μια διαφορετική προοπτική. Και θα ήταν ένα πολύ καλό μήνυμα αυτό που θα καταδείχνει ε, ότι ουσιώδη στοιχεία της συνεργασίας μας, δηλαδή μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών, μπορούν να συνεπιληθούν, να επιληθούν από κοινού. Μια τέτοια προσέγγιση είναι αυτή που προωθήθηκε και τονώθηκε από τον κύριο Καρύμ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Και δεν ήταν του κάκου, δεν ήταν μάταιη αυτή η προσέγγιση. Μια τέτοια συνεκτική προσέγγιση μπορεί να μας ε, αναγκάσει να υιοθετήσουμε μια κοινοτική επιτέλους προσέγγιση και μπορεί να μας βοηθήσει να αποφύγουμε γραφειοκρατική επιβάρυνση. Και είναι κάτι το οποίο δεν επιθυμούμε αυτή η γραφειοκρατική επιβάρυνση. Φυσικά θα κατατεθούν από πλευράς μας τροπολογίες για αυτή την έκθεση και ευελπιστούμε ότι θα εμπλουτιστεί το κείμενο της έκθεσης με αυτόν τον τρόπο και θα γίνει πιο περιεκτικό για όσους το αναμένουν. Ευχαριστώ. Κύριε Ντελβού, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ναι, και εγώ ε, πραγματικά ε, θαυμάζω τον κύριο Καρύμ για την επιμονή του. Είναι η δεύτερη φορά που παρακολουθώ την ετήσια έκθεση για την επικουρικότητα και αναγνωρίζω ότι επιχειρηματολογείται πάντα ε, προς την ίδια κατεύθυνση οπότε δεν θα εκπλαγείτε αν ακούσετε ότι εγώ δεν συμμερίζομαι την απόψή σας. Ε, εκπλήσωμαι μάλιστα διαβάζοντας έτσι λεπτομερώς την έκθεση ε, βλέπω ας πούμε ότι λέτε ότι η επικουρικότητα και η αναλογικότητα είναι οι διευθύνουσες αρχές της δράσης της Ένωσης. Αυτό με εκπλήσει δεν νομίζω να είναι οι διευθύνουσες ε, αρχές της δράσης της Ένωσης. Η Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη, στην ενισχυμένη συνεργασία, βεβαίως πάντα ε, με τη δική της ασφαλείας, της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Δεν συμμερίζομαι επίσης την ιδέα σύμφωνα με την οποία η επικουρικότητα είναι ένας τρόπος να μειωθεί το δημοκρατικό έλλειμμα. Άλλα μέσα είναι που χρειάζονται εδώ. Χρειάζονται άλλες πεπιθήσεις ε, για να μειωθεί ο ευρωσκεπτικισμός. Υπάρχει έλλειψη αλληλεγγύης, υπάρχει έλλειψη πάθους, εάν θέλετε, έλλειψη πολιτικής βούλησης σε εθνικό επίπεδο υπέρ των ευρωπαϊκών πολιτικών. Και αυτό εξηγεί τον ευρωσκεπτικισμό. Και βεβαίως λυπάμαι γι' αυτό. Επίσης δεν συμφωνώ όταν λέτε ότι πρέπει οι αποφάσεις να παίρνουν, να παίρνουν πιο κοντά στον πολίτη. Έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ τα πράγματα, εντάξει δεν είμαι βέβαιος ε, καινούργια στην πολιτική, αλλά εγώ έχω μάθει ότι οι αποφάσεις πρέπει να παίρνουν στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Σεβόμενοι την αποτελεσματικότητα της δράσης της Ένωσης και ταυτόχρονα βρισκόμενοι κοντά στον πολίτη. Δυσκολεύομαι λοιπόν να συμφωνήσω με την αρχική σας προσέγγιση. Θα υποβάλουμε τροπολογίες, εφόσον τουλάχιστον να μπορούμε να τα βρούμε για να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση διέπει και άλλες αρχές και όχι μόνο η επικουρικότητα. Η επικουρικότητα είναι ένας τρόπος για να παρθούν οι αποφάσεις στο κατάλληλο επίπεδο. Επίσης το να προσθέσουμε τώρα κόκκινες κάρτες, πράσινες κάρτες, πορτογαλί κάρτες, κάπου θα χαθούμε με τις κάρτες νομίζω. Δεν νομίζω να είναι αυτή η καλύτερη λύση έτσι ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να μπορέσουν να συμμετάσχουν και μάλιστα εκπλήσωμε. Νομίζω πως είμαστε το μόνο κοινοβούλιο στον κόσμο που θέλει να περιορίσει τις δικές του αρμοδιότητες. Δεν έχω μακρά εμπειρία κοινοβουλευτισμού, αλλά διαπιστώνω ότι αφενός ε, διεκδικούμε περισσότερη εξουσία, περισσότερε αρμοδιότητε από την Κομισιόν και το Συμβούλιο και από την άλλη δίνουμε αρμοδιότητε στα εθνικά κοινοβούλια για να μειώσουμε τα δικά μας μέσα αντίδρασης. Αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε ε, σε βάθος. Αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση εκ μέρου μου και βεβαίω αναμένω να έχουμε ε, συζητήσεις επικοδομητικέ με τον κύριο Καρύμ, του οποίου βεβαίω σέβομαι τι πεπιθήσει ε, και την αυστηρότητα των πεπιθήσεων αυτών. Παρακαλώ. Ο κύριος Λεμπρετών, να απαντήσω πολύ σύντομα στην κυρία Ντελβό, διότι άνοιξε μια συζήτηση επί της ουσίας. Ναι, είναι σημαντικό το θέμα που θίξατε. Λέτε ότι η αρχή τη επικουρικότητα δεν είναι μια κατευθυντήρια αρχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όμω το άρθρο 5 για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει έναν εξέχοντα ρόλο σε αυτή την αρχή. Κατ' εμέ λοιπόν είναι κατευθυντήρια γραμμή. Δεν είναι η μόνη, αλλά είναι σίγουρα από τι βασικέ. Τα κείμενα το λένε. Δεν μπορούμε να τα παραγνωρίζουμε σε τέτοιο βαθμό. Επίσης, μας εξηγείτε πώς δημιουργείται ευρωσκεπτικισμός. Να μου επιτρέψετε να είμαι περισσότερο εμπειρογνώμων από εσά από του θέματος, γιατί είμαι ο ίδιος ευρωσκεπτικιστής. Ξέρω πώς γίνεται αυτό και ξέρω πώς καταφέρνει κανεί να γίνει πραγματικά επιφυλακτικό προς την Ευρώπη. Όχι, δεν είναι θέμα ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έλλειψη αυτή. Είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εθνική πολιτική. Και αν θέλετε οπωσδήποτε να, και αν θέλετε να κρατήσετε και να έχετε μια μικρή πιθανότητα να σώσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή είναι ακριβώς την αρχή της επικουρικότητας θα πρέπει να ξαναδείτε. Και ίσως να ακούτε λίγο περισσότερο τι λέει ο κύριος Καρύμ. Ε, ίσως πριν φύγει μια από τις τελευταίες του προσφορές προς εσάς θα ήταν να σας κάνει να καταλάβετε πώς μπορείτε να βρείτε τρόπο να σώσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εγώ έτσι κι αλλιώ δεν είμαι υπέρ, είμαι ένας ε, σαφής πολέμιος της Ευρωπαϊκής Ένωση. Κύριε Αντελβό, απαντήστε. Με συγχωρείτε, δεν με εκπλήσει να λέτε ότι είστε ευρωσκεπτικιστής. Δεν είναι καμιά είδηση. Οπότε ναι, να συζητήσουμε. Πιστεύω ότι θα έχουμε ξανά τη συζήτηση Απλώς για την αρχή της επικουρικότητας να ξεκαθαρίσω ότι καταλαβαίνω, καταλαβαίνω ότι είναι μία από τις βασικές αρχές. Όμως αν διαβάσουμε το πρώτο εδάφιο της έκθεσης λέγεται ότι η αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας είναι οι κατευθυντήριες αρχές της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, με συγχωρείτε, αλλά είναι μία δήλωση με την οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω έτσι ως έχει. Δεν θα παραγνωρίσω την αρχή της αναλογικότητας, της επικουρικότητας, αλλά να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στη λειτουργία της κατευθύνεται από την επικουρικότητα και την αναλογικότητα αναλογικότητα κατεξοχήν είναι μια δήλωση που δεν είναι καθόλου αληθινή. Και εγώ γνωρίζω καλά τα κείμενα. Ε, άλλες παρεμβάσεις, κύριε Καρύμ, μπορείτε να ολοκληρώσετε αν θέλετε. Προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών 11 Οκτωβρίου το βράδυ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που θυμήσατε και την ε, προθεσμία για τις τοπολογίες. Προφανώς, εδώ υπάρχει μια ευρύτατη πολιτική συζήτηση που ε, αφορά αυτό το θέμα το οποίο έχω αναλάβει εδώ και χρόνια κιόλα. Να ευχαριστήσω όλου του αδέλφου για τι παρατηρήσει του ε, και όλο ιδιαίτερα τον Ταντέο που θυμίζει για πόσα χρόνια επιμελώς και συστηματικός ε, προσπαθώ να καθορίσω μία ρότα για την όλη αυτή έκθεση. Η ρότα αυτή, αυτός ο, αυτή η περιήγηση σκοπό έχει να δείξει πώς γίνεται αντιληπτή η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα κράτη-μέλη μας. Είχαμε, πιστεύω, κάποια επιτυχημένα βήματα με μερικές από τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε μέσα στα χρόνια. Κάποιοι συνάδελφοι όπως είπε ο Δαντέος, εκείνος ο ίδιος, η Αγγέλικα Νίμπλερ και άλλοι, επιβεβαίωσαν ότι ο προσανατολισμός μας ήταν σωστός. Δεν θα ήθελα τώρα να εμπλακώ κι εγώ στη σημερινή ανταλλαγή απόψεων που μόλις είχαμε. Ε, απλώς να πω ότι πιστεύω η εκθέση βασίζεται επαρκώς στα όσα προηγουμένως έχουμε κάνει. Ε, τα αισθήματά μας παραμένουν τα ίδια Αλλά σε σχέση με τις προηγούμενες συζητήσεις μας θα αισθανθώ πολύ πιο ελεύθερος να εκφραστώ για τα θέματα αυτά και βλέπω ότι, σημειώνω τι λέει η κυρία Ντελβό, σημειώνω το πολιτικό πλαίσιο που επισημαίνεται, νομίζω ότι συνεισφέρεται και εμπλουτίζεται την όλη πρόπτικη Το μόνο σχόλιο στο οποίο θα παρεκκλίνω σε σχέση με όσα υπόθηκαν είναι αυτό του κυρίου Λεμπρετών πίσω μου. Δηλαδή, νομίζω η τελευταία προσφορά μου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ασχέτως του που θα βρίσκομαι, ελπίζω να μην είναι αυτή. Οι ευχές μου και οι καλές μου ε, αναμνήσεις θα είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεισφέρω με όποιο τρόπο μπορώ στην συνέχιση της οικοδόμησής της. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, ευχαριστώ και για την τελευταία σας φράση, την ακροτελεύτια, ένα σχόλιο ε, για το οποίο κανείς εδώ, οι περισσότεροι δεν έχουμε καμία αμφιβολία, δεδομένου του πόσο χρόνο έχετε αφιερώσει σε αυτό το υπηρετικό ε, σχέδιο ένωσης για την Ευρώπη παρά τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν ξεχνάω τη θέση σας προς το Σέγγεν και καταλαβαίνω ότι αυτή σας παρέμβαση δεν είναι και αποχαιρετιστήρια, αλλά σε κάθε περίπτωση θα σεβαστούμε το έργο σας συνολικά καθώς και το πρόσωπό σας. Ε, σας ευχαριστώ. Παρεμβάσεις. Ωραία. Περνάμε στο επόμενο σημείο της μέρης διάταξης, το οποίο αφορά την έκθεση Kaufmann. Σας ευχαριστώ θέμα Πρόεδρε. Έχει προχωρήσει ο χρόνος και θα είμαι σύντομη. Είναι μια γνωμοδότηση για μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας της Επιτροπής Ελέγχου Προεκολογισμού. Πρόκειται για τον έλεγχο του Μητρώου <clears throat> και τη σύνθεση ε, ομάδων επαϊόντων πραγματογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συζητήσεις ε, για τις διαδικασίες ε, όσον αφορά τον κύριο Ντεγιόν, την κυρία Τρούιπερ και σε σχέση με την Επιτροπή Προϋπολογισμού σε διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που νέες οριζόντιες ε, διατάξεις ε, κατέθεσε που προβλέπει τις, προβλέπουν τις διαδικασίες αυτών των ομάδων πραγματογνωμόνων. Θα είμαι σύντομη και σε σχέση με την έκθεση του κυρίου Ντεγιόν για την επιλογή εκείνων των σημείων που πρέπει να εξειδικευθούν ή να συμπληρωθούν περαιτέρω. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο τρεις, ε, τρία σημεία. Το ένα είναι το θέμα της σύνθεσης των ομάδων πραγματογνωμόνων σε σχέση με τις συζητήσεις μας για αυτό το θέμα τον Ιούλιο από πλευρά συναδέλφου αναφέρθηκε ότι η πείρα και οι ικανότητες δεν πρέπει να αμφισβητούνται και αυτό το έχω συμπεριλάβει στις προτάσεις. Πιστεύω ως δεύτερο σημείο πρέπει να αναφέρουμε την ισορροπημένη σύνθεση σε σχέση με τους πραγματογνώμονες αυτών των ομάδων, ιδιαίτερα σε σχέση με οικονομικά και μη οικονομικά θέματα και συμφέροντα ώστε να υπάρχει μια ισορροπημένη ε, εκπροσώπηση, ιδιαίτερα και όσον αφορά υποεκπροσωπούμενες ομάδες, για παράδειγμα μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, ε, να μην υπάρξει εδώ κάποια απουσία ή ε, έλλειψη χρηματοοικονομικής ε, υποστήριξης, συνδρομής. Είναι σημαντικό εδώ να ε, δίνει τα εγχέγγυα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ταυτόχρονη διαβίβαση αυτών των στοιχείων για τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις και φυσικά είναι αυτονόητο ότι για αυτές τις πράξεις δυστυχώς δεν είναι πλήρη τα στοιχεία και ως εισηγήτρια θα ήθελα να καταθέσω μια τροπολογία επ' αυτού ώστε να ενταχθεί και αυτό το σημείο και περαιτέρω θα συζητήσουμε και ελπίζω ότι οι συνάδελφοι θα μπορέσουν αυτή τη γνωμοδότηση να την προαγάγουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για την παρουσίαση που δόθηκε. Καλύπτει πολλά στοιχεία και είναι σημαντικό εδώ να μπορέσουμε για αυτό το θέμα να δράσουμε όπως πρέπει γνωρίζοντας ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο δραστηριοποιούν τέτοιες ομάδες πραγματογνωμόνων και πρέπει να διασφαλίσετε ότι θα υπάρχει διαφάνεια και για τη σύνθεση αυτών των ομάδων έχει γίνει συζήτηση ήδη σε σχέση με την Επιτροπή και για θέματα αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων. Χρειαζόμαστε μια ισορροπημένη εκπροσώπηση και σύνθεση σε αυτές τις ομάδες και γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει αυτές τις προτάσεις. Τονίζω για άλλη μια φορά ότι είναι ουσιώδες Συμβούλιο και Επιτροπή να συγκαλούν τέτοιους πραγματογνώμονες που θα έχουν πείρα και θα είναι ε, πέρα από πεπειραμένοι, θα είναι και αποτελεσματικοί. Συχνά για προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν υπάρξει εκτενείς συζητήσεις για προτάσεις πραγματογνωμόνων που δεν είχαν όμως πείρα. Και αναφέρομαι σε σχέση με την Επιτροπή Οικονομικών και μπορώ εδώ να το αναφέρω αυτό και να τονίσω ότι υπάρχουν τέτοιου είδους ομάδες πραγματογνωμόνων που όταν συγκαλούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Συμβούλιο πρέπει να έχουν τις ικανότητες και την πείρα που χρειάζονται. Μάλιστα, δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Ωραία, πάμε στο επόμενο σημείο της διάταξης που είναι η έκθεση του κυρίου Γέσικα. Le rapport de Η έκθεση του κυρίου Σβόμποντα, πιο συγκεκριμένα, την οποία όμως μας παρουσίασε, παρουσίασε εδώ ο κύριος Βιέτσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ακριβώς γι' αυτόν εδώ τον λόγο, πραγματικά, που από πλευράς του κυρίου Σβόμποντα που α, ε, δεν μπορεί να παραστεί, αλλά θα, μπορεί να, θα μπορέσει να επανέλθει ευελπιστούμε σύντομα. Μου ζήτησε να παρουσιάσω, να εκθέσω εγώ τις αλλαγές όσον αφορά τους κανονισμούς, τον, ε, τον κανονισμό του Ευρωκοινοβουλίου. Αφορά ένα έγγραφο το οποίο από ειδική επιτροπή συντάχθηκε μέσα στο, στους κόλπους της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Υπάρχουν όμως σημαντικές αμφιβολίες όσον αφορά τις αποκλειστικές αρμοδιότητες αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και αυτό θα πρέπει να τονιστεί και σε σχέση με το έγγραφο του εισηγητού και υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να τονίσουμε εδώ όσον αφορά για παράδειγμα ασυλίες και θέματα που αφορούν νομικές βάσεις Μπορεί να ενθυμίστε ότι αυτά τα θέματα κατά το παρελθόν ε, υπάρχουν και δείχνουν ότι οι διαδικασίες θα μπορούσαν να ε, βραχυνθούν, να συντμηθούν σημαντικά και ίσως ε, με την εγκατάλειψη των διαδικασιών ε, ψηφοφοριών σε σχέση με άρση ασυλιών. Η ιδέα είναι ότι θα έπρεπε η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων να επιλαμβάνεται αυτών των ε, ζητημάτων και όσον αφορά τα αιτήματα των ενδιαφερομένων θα μπορούσαν ίσως ε, αυτά να ψηφίζονται στην Ολομέλεια. Ε, δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί το θέμα των, προτάσεων των συντονιστών. Πρέπει να διατηρηθεί η υφιστάμενη διαδικασία η οποία λειτουργήσε επί ολόκληρη σειρά ετών. Θα ήταν πολύ δύσκολο να εξευρεθεί μια καλύτερη λύση διαδικαστικά. Για τα άλλα θέματα τα οποία τίθενται υπό συζήτηση όπως τη νομική βάση για παράδειγμα οι τροπολογίες οι οποίες αφορούν για παράδειγμα τη νέα διοργανική συμφωνία το κείμενο της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων σαφώς καταδεικνύει ότι υπάρχουν κάποιοι λανθασμένοι προσανατολισμοί σε κάποια ζητήματα και για τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται και σε σχέση με το έγγραφο της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και την δέσμευση άλλων θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις εσωτερικές διαδικασίες που ακολουθούν από αυτά. Είναι μια, θα έλεγα, παράλογη όμως λύση αυτή, διότι το συγκεκριμένο αυτό έγγραφο αφορά αποκλειστικά μόνο τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εδώ εξαπίνεις προτείνουμε λύσεις ε, για άλλα θεσμικά όργανα. Αυτό είναι απαράδεκτο, Πρόεδρε. Και αυτό θα μπορούσε να προσβληθεί, να υποστεί οποιαδήποτε αμφισβήτηση από οποιονδήποτε. Άλλες ε, τώρα προσεγγίσεις που χρειάζονται, που χρήζουν αποσαφηνήσεων όσον αφορά ε, τις διαδικασίες, όσον αφορά την επικουρικότητα, την κατεξουσιοδότηση πράξης, ε, για παράδειγμα, όσον αφορά επίσης αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα σε σχέση με το άρθρο 5, το 256 σε σχέση με διεθνείς συμφωνίες και νομοθετικές πράξεις μεταξύ άλλων. Αυτά ίσως τα σημεία δεν είναι εξίσου κατεπήγοντα και θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι θα μπορούσαν να ε, εξεταστούν εν ευθέτω χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κάφμαν, έχεις στο λόγο. Η κυρία Κάφμαν, σας ευχαριστώ θερμά πρόεδρε και ευχαριστώ επίσης και τον κύριο Σβιεύκα για την παρουσίαση. Θέλω μόνο σε δύο σημεία να πω δύο λόγια. Το πρώτο είναι το θέμα των διαδικασιών ασύλειων. Ο συνάδελφος Βιεύκα ε, διεξοδικά τοποθετήθηκε από αυτού. Θεωρώ πράγματι ότι είναι σημαντικό να παραμείνουμε στις διαδικασίες όσες έχουν και εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή. Μια συστηματική ψηφοφορία για κάθε αίτηση άσης ασυλίας στην Ολομέλεια απαιτείται και τώρα το γιατί επιθυμούν κάποιοι να τροποποιήσουν αυτές τις διαδικασίες δεν μπορώ να το κατανοήσω. Για θέματα νομικής ασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντικό να διεξάγονται τέτοιου είδους ψηφοφορίες όταν υπάρχουν τέτοια αιτήματα. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο οπωσδήποτε ήθελα να υπογραμμίσω. Για την άλλη μου παρατήρηση ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Σβέφκα να διαβιβάσει στον κύριο Σβόμποντα ως εισηγητή ότι έχουμε σημαντικές επιφυλάξεις επί ενός σημείου. Και θεωρούμε ότι εδώ δημιουργείται μια κατάσταση τουλάχιστον όπου θεωρώ ότι η πλειοψηφία της ομάδας μου δεν μπορεί να υπερψηφίσει. Πρόκειται για μια πρόταση να τροποποιηθεί η διαδικασία όσον αφορά την επικουρικότητα στην Ευρωβουλή και προτάθηκε το άρθρο 42 να τύχει μιας νέας υποπαραγράφου, ενός νέου υποεδαφείου, ένα, ενός 1α. Είχαμε τη συζήτηση για την επικουρικότητα με τον κύριο Κάριμ και πιστεύω ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων είμαστε υπερήφανα για την αρμοδιότητα αυτή που έχουμε για την εξέταση θεμάτων επικουρικότητας στην Ευρωβουλή. Έχουμε μια πρόταση τώρα από τον συνάδελφο Σβόμποντα που πιστεύω ότι αποδυναμώνει σημαντικά τις αρμοδιότητές μας ως μελών της ε, ε, Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και δίνει μια δυνατότητα όλες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές εξίσου να έχουν αρμοδιότητες και να εξετάζουν θέματα επικουρικότητας εναλλάξ και αυτή, αυτή η εξέταση να ανακυκλώνεται σε διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές και να υπάρχει έτσι, ας το, ας το αποκαλέσω έτσι, αυτοαπασχόληση για να έχουν κάτι να κάνουν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές. Αυτό όμως δεν είναι καθόλου συμβατό με τις αρμοδιότητες τις δικές μας και των άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Όχι μόνο αυτό ε, θα πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά, αλλά να, όταν ζητηθεί αυτό από κάποιους ευρωβουλευτές και ακολουθηθεί αυτή η διαφορετική διαδικασία θα προκληθεί χάος. Πρέπει να παραμείνουμε σε αυτή τη διαδικασία σε σχέση με το άρθρο 42 εδάφιο 2 ως έχει και να μην τροποποιηθεί. Ευχαριστώ θερμά. Merci beaucoup, madame. Pas Ευχαριστώ. Δεν φαίνεται θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Πολύ ωραία. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο τη ημέρα διάταξη. Η κυρία Κομοντίνη Λύπη. Λοιπόν, το επόμενο σημείο είναι το θέμα της νομικής βάσης. Στην προηγούμενη συνάντησή μας μιλήσαμε για το θέμα της νομικής βάσης της πρότασης κανονισμού για τη δημιουργία ενός οργάνου συνεισφοράς στην σταθερότητα και την ειρήνη. Αυτή η δεύτερη αλλαγή απόψε ελπίζω να βοηθήσει τους συναδέλφους που έχουν ακόμα δισταγμού να μπορέσουν να διαμορφώσουν μια σαφή θέση για το θέμα. Εγώ προσωπικά είμαι πεπισμένος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιλέξει την κατάλληλη νομική βάση. Δηλαδή και συνεργασία για την ανάπτυξη και τεχνική και οικονομική συνεργασία. Όπως σας πρότεινα την προηγούμενη φορά, ο γενικός στόχος της πρότασης είναι να, προστατεύονται οι πολίτες σε ζώνες σειράξεων ή στα πλαίσια μιας δύσκολης πολιτικής συγκυρίας που ε, διακινδυνεύει όπου διακινδυνεύουν οι πολίτες ε, την ασφάλειά τους, λαμβάνοντας βέβαια πάντα υπόψη και την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική προστασία στις χώρες αυτές. Ε, το στρατηγικό σκέλος του εγχειρήματο πρέπει να εγγραφεί ε, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αυτός ο εξαιρετικός χαρακτήρας της στρατιωτικής συνδρομής δείχνει ότι αυτή η συνιστόσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως ίστατη λύση. Η μόνη αποδεκτή αιτιολόγηση είναι σοβαρή απειλή στους θεσμούς μιας χώρας ή των, των θεμελιών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του πληθυσμού της. Όταν δηλαδή οι θεσμοί της χώρας αυτής δεν μπορούν πια να κάνουν τίποτα. Η συνεργασία για την ανάπτυξη πολύ μικρή ε, επιρροή μπορεί να έχει αν δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι λοιπόν προφανές ότι αυτή η πτυχή τη στρατιωτική συνδρομής πρέπει να προβλεφθεί. Πρέπει να έχετε να καλύψει, να συμπληρώσει την αρχική κάλυψη. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η πρόταση απαγορεύει να χρησιμοποιηθεί αυτό το μέσο για την χρηματοδότηση ε, στρατιωτικής εκπαίδευσης, ε, την τη χρηματοδότηση της, ε, του, του ανεφοδιασμού σε όπλα ή σε πυρομαχικά. Ε, έτσι λοιπόν δεν μπαίνει εδώ ζήτημα σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι αυτά είναι και τα βασικά επιχειρήματα που πρέπει να λάβει υπόψη της η Επιτροπή μας. Από εκεί και πέρα η αρμόδια επιτροπή ε, θα αποφασίσει επί της ουσίας για τη σκοπιμότητα ενός τέτοιου μέσου ε, και υπό ποιες προϋποθέσεις βέβαια θα μπορούσε να υπάρξει. Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας η αρμόδια επιτροπή λίγο πολύ αυτή τη γραμμή την οποία σας περιέγραψα ακολουθεί αυτά που σα είπα και την προηγούμενη φορά δηλαδή. Όμω επειδή υπήρξε αυτό το αίτημα εξέταση τη νομική βάση, ε, θα αναφερθώ εγώ στους πολιτικούς λόγους για τους οποίους ε, θεωρούμε εμείς σκόπιμο να παραμείνει η νομική βάση. για να διατηρήσουμε την παρούσα νομική βάση, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι η σύνηθις νομοθετική διαδικασία που επιτρέπει στους Ευρωπαίους βουλευτές να εξασφαλίσουν ότι θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί αυτό το μέσο ε, για τον σωστό σκοπό και για ανθρωπιστικούς λόγους. Εμείς είμαστε υπέρ μιας πολιτικής ασφάλειας, κοινή ασφάλειας, κοινή άμυνας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν και το δικαστήριο ε, θα μείνουν εκτό αν ακολουθηθεί αυτή η πολιτική ασφάλειας και άμυνας, ακολουθεί αυτό ο πυλώνας. Τότε δεν θα έχουμε πια λόγο αν αλλάξουμε δηλαδή, την νομική βάση. Να σας πω επίση επίσης ότι μέρος του προπολογισμού αυτής της πολιτικής προέρχεται απευθεία από τα κράτη-μέλη και οι αποφάσεις παίρνονται ομόφωνα μόνο από το Συμβούλιο. Κάποιοι συνάδελφοί μου είπαν ότι θα ήθελαν να ακούσουν την άποψη της νομικής υπηρεσίας της Κομισιόν και του Συμβουλίου για, το, για την καταλληλότητα της νομικής βάσης. Αναμένοντας μια γραπτή απάντηση εκ μέρους τους, μπορώ να καλέσω τους εκπροσώπους των οργάνων αυτών να μας πούν την άποψή τους. Θα ήθελα δηλαδή, ιδιαίτερα να ακούσω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας πει δηλαδή ποια είναι τα επιχειρήματα ε, ποιοι είναι οι λόγοι που έγινε αυτή η επιλογή, κατά πόσο αυτή η επιλογή είναι κρίσιμη σημασίας ε, και για μελλοντικά παρεμφερεί με νομοθετικά μέσα. Αυτά είχα να πω. Αναμένω τώρα τα σχόλιά σας, τα ενδεχόμενα σχόλιά σας. Η κυρία Ράινερ. Ευχαριστώ θερμά κύριε Πρόεδρε για αυτά που μας αναφέρατε μόλις τώρα και που είναι εύλογα. Ευχαριστούμε πολύ για το έργο και για τα επιχειρήματα αυτά. Παρ' όλα αυτά όμως θα ήθελα κάποια επιχειρήματα να παρουσιάσω και να πω να έχουμε κάποια περισσότερη υπομονή και σε σχέση με τη σκιώδη εισηγήτρια που είναι αρμόδια για αυτό το θέμα και έχουμε εδώ και το θέμα μικροφορολογουμένων και που δεν είναι δυνατόν σήμερα να ε, παρουσιαστεί. Είναι ένα θέμα λοιπόν που καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια γι' αυτό και σε σχέση με τους σοσιαδημοκράτες δημιουργήθηκε και μια ομάδα εργασίας. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, δεν είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την κατάσταση αυτή. Προσπαθούμε όμως να έχουμε μια ένα καλό επιχείρημα που θα μπορεί να τεκμηριώνεται νομικά με τα ε, νομικά εκείνα στοιχεία που θα επαρκέσουν θα πρέπει να μπορέσουμε αυτά τα επιχειρήματα να λάβουμε υπόψη συνιστώ να έχουμε λίγη, υπομονή, λίγη μεγαλύτερη υπομονή ώστε να μπορέσουμε σε σχέση με το θέμα αυτό να προχωρήσουμε λίγο και να συζητήσουμε με, τους, ε, με τα αρμόδια μέλη Έχουμε λοιπόν πραγματικά ε, ένα θέμα το οποίο είναι ακαθόδες ε, και φλέγον πολιτικά. Λοιπόν, κοντός ψαλμός αλληλούια. Λίγη υπομονή λοιπόν παρακαλώ μέχρι να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Αναντήρητα. Τα κατεπήγοντα μπορούν να περιμένουν. Ε, γι' αυτό και ο Σιώδης εισηγητής δεν είναι εδώ από την ομάδα σας. Ε, κάποιος θέλει το λόγο για το θέμα αυτό, κύριο Σιεφκά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης του ΕΛΚ για αυτό το θέμα και ήθελα να συμμεριστώ την επιχειρηματολογία σας ως εισηγητού. Ναι, πράγματι πρόκειται για ένα ζήτημα σοβαρών ίσως όχι τόσο περίπλοκο όσο μερικοί προσπαθούν να μας παραστήσουν, όμως πρέπει να το εξετάσουμε με, τον δέοντα, ε, με τη δέουσα προσοχή. Και όταν ληφθεί η ανάλογη απόφαση θα πρέπει να ληφθεί τεκμεριωμένα για να έχουμε λάβει υπόψη τις απόψεις όλων όσοι ασχολούνται με το θέμα. Ακούγονται κάποιοι φόβοι ότι η νομική βάση για την πολιτική ανάπτυξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άλοθη για να προβλεφθούν ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις στις ε, οικίες χώρες. Δεν ισχύει αυτό, είναι τελείως και θα πρέπει να το αντικρούμε. Ε, επίσης, ο κ. Καβαντά μας απέδειξε ότι το εργαλείο αυτό θα είναι πολύ αποτελεσματικό όταν προσπαθούμε να επιλύσουμε συγκρούσεις ή για την πρόληψη τέτοιων. Παρόμοιες απόψεις ακούμε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Πιστεύω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά μαζί. Ας περιμένουμε Ας περιμένουμε τις απόψεις των υπόλοιπων συναδέλφων και θα αποφασίσουμε μετά. Ευχαριστώ. Προφανώ, προφανώς θα περιμένουμε να συγκεντρωθούν όλε αυτέ τι απόψει, ώστε να είναι ε, πολιτικά ακλόνητο το κείμενο αυτό. Ε, υπάρχουν άλλε απόψει, συνάδελφοι. Όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει πολύ γρήγορα να πει την άποψή τη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζαν Λουίφη, είμαι ε, υπεύθυνο τη Γενική Διεύθυνση, με τη της στη Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ. Άκουσα την εκκλησία σα, καθώ και αυτό που είπατε για την ανάγκη να ε, υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των νομικών μα υπηρεσιών, ιδίω αυτή τη Επιτροπή. Φαντάζομαι ότι δεν λάβατε την απάντησή μας. Απάντηση που η νομική υπηρεσία της Επιτροπής συνέταξε ε, εξ ονόματος του Γενικού Διευθυντή την Παρασκευή. Δυστυχώς δεν έχει φτάσει σήμερα από ό,τι φαίνεται. Εκεί εξηγούμε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη άποψη ε, καταγεγραμμένη για αυτήν την πρόταση. Επιβεβαιώνεται όμω έτσι ότι η νομική υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχε σε όλε τι προπαρασκευαστικέ φάσει για την εκπόνηση αυτή τη θέση. Μαζί μου είναι η συνάδελφος Αλεξάνδρα Μπαρτέλη, η οποία ε, είναι από την νομική υπηρεσία και μπορεί προφορικώς να σας δώσει κάποιες διευκρινήσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η δική σας η μελέτη του θέματος. Εάν συμφωνείτε θα της δώσω λοιπόν το λόγο. Σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ε, σωστά ε, επισημάνατε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρότεινε τροποποίηση για το εργαλείο που έχει σκοπό να συνεισφέρει στην ειρήνη και την ανάπτυξη, διευκρινίζοντας υποποιούς όρους η στήριξη των φορέων ειρήνης συμπεριλαμβανομένων των δράσεων θα μπορούν να λάβουν χώρα βάσει του άρθρου 209 και 212 για την ε, γενικότερη συνδρομή τη ε, χώρα εταίρου. Η πρόταση αυτή έχει προχωρήσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει την πλήρη στήριξη τη νομική υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει παρακολουθήσει στενά τη σύνταξη τη εν λόγω πρόταση και στηρίζει την επιλογή αυτή τη νομική βάση, όπω υπόθηκε και στο προήμιο αυτή, καθώ και στο νομοθετικό κείμενο το ίδιο, στο σώμα του κειμένου. Ε, τώρα να στραφώ στο θέμα της ίδιας της νομικής της βάσης. Προκύπτει από την αρχή της χώρισης ε, αρμοδιοτήτων, ε, εξουσιών και έχει γίνει η χώρηση αυτή βάσει της σωστής νομικής βάσης για το πεδίο της αναπτυξιακής συνεργασίας, όπως ερμηνεύτηκε και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και όπως αντικατοπτρίζεται στο δικό σας σημείο κύριε Σιγητά. Θεωρούμε ότι η χρηματοδότηση διοικοδόμησης δυνατοτήτων στον τομέα ασφάλειας και βάσει των άρθρων 209 και 212 ε, βάσει των προϋποθέσεων της πρόθεσης δεν μπορούν αυτές καθεαυτές να αποκλείονται μόνον και μόνον λόγω της θετικής φύσης ε, του δικαιούχου. Ε, διαφωνώ, διαφωνώντας να πω ότι δεν προβλέπεται στην, αναπτυξιακή, στην, στην πολιτική αναπτυξιακή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κανένα πρόβλημα δηλαδή πολιτική οικοδόμηση και στρατιωτικές δράσεις στα πλαίσια της ε, ε, κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνας κατά παραβίαση του άρθρου 40. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της πρότασή μας. Ε, το κέντρο βαρύτητας της πρόταση πρέπει να λάβει υπόψη ιδίω σοβαρότατε εξελίξει στο διεθνέ προσκήνιο που έχουν ενεργοποιήσει και την όλη μα πρόταση. Από τη μια η έγκριση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξη και από την άλλη η αναθεώρηση παλαιότερων οδηγιών στα πλαίσια της ειρήνης και τη ασφάλεια Κάποιε σαφεί ενδείξει για το κατά πόσον και υπό ποιου όρου είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ε, χωρών εταίρων. Είναι σαφές ότι το πεδίο τη αναπτυξιακή συνεργασία τη Ευρωπαϊκής Ένωση δεν συμπίπτει πλήρω με την ε, ε, στρατιωτική στήριξη που προκύπτει από την πολιτική άμυνας αλλά δεν μπορούμε να βγούμε εκτός και αυτού του πεδίου τελείως, πέραν από έκτακτε συνθήκες, όπως εκεί όπου έχουν γίνει δυσλειτουργικές για την παροχή βασικών υπηρεσιών ε, οι θεσμικές δομές ενός κράτους και για την εύρυθμη λειτουργία μιας κοινωνίας. Δηλαδή η εύρυθμη λειτουργία τους δεν μπορεί να εξασφαλιστεί από τις πολιτικές αρχές. Υπ' αυτές τις συνθήκες θεωρούμε δυνατό να ξεπεράσουμε τόσο προβλέπει η ODA η αναπτυξιακή συνεργασία δηλαδή, να παράσχουμε και στρατιωτική στήριξη, όπως ε, διευθυνίζουν και αναφερειμένες οδηγίες. Θεωρούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η ανάπτυξη της χώρας που ε, συζητούμε μπορεί μόνο στρατιωτικά να ε, προχωρήσει και με την ανάγκη οικονομική στήριξη προκειμένου να αποκατασταθεί το κράτος δικαίου στην λόγω χώρα, τη χώρα εταίρο. Η φύση των δράσεων υπερισχύει των ίδιο των δράσεων. Υπ' αυτέ τι έκτακτε ε, προποθέσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα περίπτωση εξέταση για να δούμε κατά πόσο πληρούνται αυτέ οι προποθέσει. Θα πρέπει να αναζητήσει σκόπιμου τρόπου ο προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνεισφέρει στη σταθερότητα των χωρών εταίρων. Βεβαίω, αυτό που δεν προβλέπεται είναι μια διεξοδική συνολική λύση για τις ε, περιπτώσεις της ε, ασφάλειας και άμυνας και της ε, κοινή πολιτικής. Ε, αυτό αναφέρεται στο ε, προήμιο, δηλαδή εάν θέλουμε τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών δράσεων για αμυντικούς σκοπούς να την επιτρέψουμε, θα πρέπει να προβλέψουμε εργαλεία εκτός του προπολογισμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να υπογραμμιστεί και ελπίζω ότι με αυτές τις διευκρινήσεις διευκόλυνα την μελέτη του όλου θέματος από πλευρά ναι, με μία μόνο διαφορά ότι πολλοί σε αυτή την αίθουσα δεν ξέρουν τι είναι το CBSD, αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε, για να καταλαβαίνουμε και τι λέμε. Ε, ε, με συγχωρείτε, συγγνώμη, είναι η στήριξη της ασφάλειας και ανάπτυξης καθώς και οικοδόμηση δυνατοτήτων. Αυτό ήταν και η αφορμή γέννησης της πρότασης, διότι όταν ξεκινήσαν οι συζητήσεις ε, στις ε, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης οδηγηθήκαμε στην δημοσίευση της κοινή μα ανακοίνωση για το θέμα αυτό, την οικοδόμηση δυνατοτήτων και την στήριξη της ανάπτυξης και προ προτάσεις για τροποποίηση του εξωτερικού χρηματοδοτικού εργαλείου. Αφού εκπονήθηκε και ζητηθήσα μελέτη αντικτύπου, στα πλαίσια αυτή τη οικοδόμηση δυνατοτήτων συνεχίσαμε τι προτάσει μα. Σα ευχαριστώ πολύ για την διευκρίνηση και σα ευχαριστώ. Δεν φαίνεται να θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Δεν χρειάζεται νομίζω να αντλήσουμε κάποιο συμπέρασμα. Είναι σαφή τα πράγματα. Είμαστε βέβαια στη διάθεση όλων όσων χρειάζονται λίγο χρόνο για να βελτιωθεί το κείμενο. Σα ευχαριστώ πολύ για τι προτάσει σα πάντω, όπω συμφωνήσαμε με τη Γραμματεία, είμαι υποχρεωμένο να ε, φύγω, διότι έχω ένα πολύ σημαντικό ραντεβού, σχεδόν τόσο σημαντικό όσο η σημερινή συνεδρίαση, οπότε η συνάδελφος θα αναλάβει την Προεδρία. Ε, ο... Από τον ένα στον άλλον περνάμε. Περνάμε στο σημείο 14. Εξέταση των κατεξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών μέτρων. Η κυρία Φεράρα απουσιάζει. Δεν είναι εδώ. Δεν έχει καμία αντίρρηση όμως, οπότε μπορούμε να το εγκρίνουμε. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτό το σημείο. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Αυτό είναι το τελευταίο σημείο για την ανοιχτή μας συνεδρίαση και τώρα ξεκινάμε την κεκλεισμένα των θυρών. Προσκαλώ όλους όσοι δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στη συνεδρίαση κεκλεισμένα των θυρών να εξέλθουν. Παρακαλώ φύγετε. Διακοπή ενός λεπτού για να φύγουν όλοι. Uh, thank you.